Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Would you please, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Oh, work. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε παρακαλώ να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. So, dear colleagues, good afternoon. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Πριν ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, να σας ενημερώσω ότι ο, ο φάκελος που συνήθως έχετε μπροστά σας ακόμα δεν έχει έρθει λόγω προβλημάτων μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ε, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει και θα σας διανεμηθεί το συντομότερο δυνατόν. Α Ας πάμε λοιπόν στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση ή κάποιες αλλαγές που θέλετε να προτείνετε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε? Ωραία, να σας θυμίσω ότι υπάρχει διερμηνία σε 16 γλώσσες. Δεν υπάρχει στα ε, δανέζικα, σουηδικά, εσθονικά, λετονικά και σλοβένικα. Uh, το νούμερο 2. Εγκρίση των πρακτικών 4η ε, Ιανουαρίου 2010 και 25 Ιανουαρίου 2010. θεωρούνται ότι εγκρίθηκαν στο τέλος της ε, συνάντησης, της ε, συνεδρίασης, εάν δεν υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις που αγευθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Το σημείο 3 θα μας ε, το παρουσιάσει αργότερα η κυρία Χούμπνερ. Και πάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, γενικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά την απλούστευση συγκεκριμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικά με την οικονομική διαχείριση. Σε αυτό το σημείο δίνω το λόγο ε, δίνω το λόγο στον εισηγητή στον κύριο Κυρίλοφ. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ε, ε, πληροφορήσω ότι η διαφωνία που υπάρχει με την Επιτροπή Απασχόλησης ε, έχει λυθεί σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνο. Οι Επιτροπές Απασχόλησης και Προϋπολογισμού θα κάνουν γνωμοδότηση στο έγγραφο της Κομισιόν. Αυτή η τελευταία διευκρίνηση της διαδικασίας μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε το σχέδιο ε, πρότασης ε, της ε, Κομισιόν για την τροποποίηση του γενικού κανονισμού. Προτείνω κάποιες τροπολογίες που θα αλλάξουν την πρόταση της Κομισιόν από τον Ιούλιο του 2010, όπως ανακοινώθηκε στις 18 Ιανουαρίου στην Ολομέλεια. Αυτές οι τροπολογίες περιλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο. Το σχέδιο ήδη έχει προταθεί και παρουσιαστεί στην Επιτροπή μας. Έχουμε το δεύτερο έγγραφο εργασία, το οποίο συζητήσαμε τον Ιανουάριο στη συνεδρίασή μας. Παρόλο που το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη από το Σεπτέμβρη, θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω τις βασικές τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν και στο σχέδιο της έκθεσης. Δεν είναι δικές μου, παρουσιάζω τις τροπολογίες της Κομισιόν και του Συμβουλίου τροπολογία της πρότασης της Κομισιόν ε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Πρώτον, σχετικά με την, ε, τους κανόνες οικονομικής διαχείρισης δημοσιονομικής διαχείρισης ε, για τα προγράμματα συγχρηματοδότησης του Κοινωνικού Ταμείου και δεύτερη ομάδα εφαρμογή των προγραμμάτων για όλα τα ταμεία. Οι τροπολογίες που προτείνονται στο σχέδιο της έκθεσης αναφέρονται και στις δύο ομάδες. Πιο σημαντικέ όμω είναι οι τροπολογίε που σχετίζονται με του κανόνες της δημοσιονομική διαχείριση. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση της περιφερειακή Επιτροπής προβλέπει μία επιλογή για τα κράτη-μέλη να λάβουν 100% επιστροφές των ενδιάμεσων πληρωμών και των απαιτήσεων που έχουν για το Κοινωνικό Ταμείο 2009-2010. Παρά το γεγονός ότι Αυτέ οι τροπολογίε του άρθρου 77 θα είναι για περιορισμένο διάστημα και η συγχρηματοδότηση θα παραμείνει ως υποχρέωση για όλη την προγραμματική περίοδο. Αυτό είχε επικριθεί από τα κράτη-μέλη, γιατί λένε ότι παραβιάζει τη βασική αρχή της κοινοτικής χρηματοδότησης ότι είναι περίπλοκη και δαπανηρή. Επίσης, ε, εδώ στις συνεδριάσεις μας υπήρχαν επικρίσεις. Συμφωνώ και ε, Υποστηρίζω την τροπολογία των άρθρων 82 και 93 για να ε, αντικαταστήσουν την τροπολογία του άρθρου 77. Επίσης, η τροπολογία σχετικά με τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση να λάβουν προκαταβολές 2% του ε, Ταμείου Συνοχής και 1% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουν ε, θεσπιστεί σε σχέση με αυτό κάποια αντικειμενικά ε, κριτήρια για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση των κρατών μελών. Τροπολογία του άρθρου 93 θα μας επιτρέψει ε, μια ευελιξία στους, ε, στις αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2007, οι οποίες θα χωριστούν σε έξι μέρη και το ένα έκτο θα προσθεθεί ε, σε κάθε έτος από το 2008 στο 2013. Έτσι θα γίνει μια σωστή ε, διανομή του οικονομικού φόρτου για το 2007 σε όλη την περίοδο και έτσι οι χώρες θα μπορέσουν ε, να ανταποκριθούν. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ καλή και χρήσιμη για όλες τις χώρες, γιατί όπως γνωρίζετε όλα τα κράτη-μέλη πήραν ε, πολύ αργά την έγκριση για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του 2007. Ως εισηγητής έχω επαναλάβει την ε, ρητή υποστήριξή μου στην πρόταση της ε, Κομισιόν για την απλούστευση των κανόνων. Στα διορθωτικά ταμεία ε, υπάρχουν μόνο κάποιες μικρές αλλαγές που έχω στο σχέδιο έκθεσης. Γενικά η πρόταση απλούστευσης ε, εμπίπτει στα εξής άρθρα του Γενικού Κανονικού, ε, Κανονισμού. 50 εκατομμύρια ευρώ ως κατόφλι για τα ε, προγράμματα και δυνατότητα χρηματοδότησης ως ενιαίο πρόγραμμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν εμπλέκονται διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτό σημαίνει μία έναν διαχωρισμό σε κάποια προγράμματα, ο οποίος ε, θα βελτιώσει τη συνοχή μεταξύ των δράσεων και θα βελτιώσει τη διαχείριση των προγραμμάτων. Επίσης, προτείνεται οι δαπάνες για μεγάλα προγράμματα να προστατεύονται από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη δέχονται, ε, υποβάλλουν την ε, πρόταση στην Κομισιόν και όχι από την έγκριση όπως γίνεται τώρα άρθρο 94 και πάλι για να εξοικονομούμε χρόνο. Πολλά μέτρα πλούστευσης επίσης προτείνονται για να ε, μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες δαπάνες ε, στην αποδοτικότητα της ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Συγκεκριμένα θέλουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο ε, το οποίο προτείνεται στο άρθρο 44 και υπάρχουν ε, και δαπάνες ε, διαχείρισης που είναι μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών άρθρο 78 και 7 σχετίζονται άμεσα με τον προηγούμενο γύρο τροποποιήσεων 2008-2009 και όλα αυτά τα άρθρα έχουν αναδρομική ισχύ από το 2009 για να διευκολύνουμε την υιοθέτηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα οικονομική κρίση, τα κράτη-μέλη δίνουν ανάλυση που δικαιολογεί την αναθεώρηση ενός επιχειρηματικού προγράμματος, άρθρο 48. Επιπλέον, δεν θα γίνει αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος, δεν χρειάζεται πλέον για όχι εντελώ καινούργιε κατηγορίε δαπανών, άρθρο 56 πιο βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ε, για την παρακολούθηση των ε, εσόδων επίσης έχουν εισαχθεί και αυτό είναι το άρθρο 55. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε το άχθος της ε, λογοδοσίας υπάρχει μια ανάγκη για αναφορά σχετικά με την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με τις αιτήσει πληρωμών κάθε έτος. Επίσης υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σχετικά με το γενικό κανόνα για τα κονδύλια που εφαρμόζονται μόνο σε υποδομές ε, παραγωγικών ε, επενδύσεων, όχι για άειλες επενδύσεις. Δεύτερον, για τη ε, διαδικασία του κοινωνικού ταμείου, κρατική ενίσχυση, η κοινοτική συνδρομή θα διατηρείται μόνο εάν υπάρχει τέτοια υποχρέωση σύμφωνα με τις κρατικούς κανόνες. Δουλεία, χρεοκοπία και ε, εξαιρούνται. 57 άρθρο. Επίσης, Όλα αυτά έχουν γίνει για να απλουστευτεί η καταβολή των προκαταβολών στους δικαιούχους και να μειωθεί ο οικονομικός κίνδυνο που σχετίζεται με αυτές τις πληρωμές. Ξεκαθαρίζεται τώρα ότι οι παραδεκτές εγγύσει δεν είναι μόνο αυτές που προέρχονται από τις τράπεζες, αλλά και από δημόσιε οντότητες ή κράτη-μέλη. Άρθρο 78 τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το μερικό κλείσιμο των προγραμμάτων περισσότερο ε, με μια νέα διάταξη η οποία λέει ότι σε περίπτωση ασυνεπιών που εντοπίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη και όχι η Όλαφ τα διορθωμένα ποσά μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα ενώ τώρα χάνονται και έτσι τα κράτη-μέλη δεν έχουν τέτοια επιλογή. Άρθρο 88 Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ μια πολύ ε, καλή ενθαρρυντική τροπολογία για τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να εμπλέκονται πιο ενεργά στον έλεγχο. Αυτές, εν συντομία, ήταν οι τροπολογίες που σας προσκάλω να υποστηρίξετε. Αυτή είναι ρεαλιστικά η τελευταία αλλαγή του γενικού κανονισμού για την ε, τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ώστε να αλλάξουμε ε, να μην αλλάζουμε συνεχώς τους κανόνες που θα κάνουν δύσκολη τη ζωή των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων. Απ' την άλλη να πω ότι Έχουν γίνει ακουστές ε, οι ανησυχίες των κρατών μελών, οι πρακτικές που γίνονται σε όλη τη διαδικασία, που χρησιμοποιούνται σε όλη τη διαδικασία Ίσως όχι όλα, αλλά συμφωνήσαμε και ο Νέος Επίτροπος επίσης ε, συμφώνησε ότι αυτή η διαδικασία θα είναι συνεχής και το ζήτησα αυτό. Επίσης λοιπόν ε, να σας πω ότι θα εκτιμάτε η μελλοντική συμβολή της Επιτροπής. Ακούσαμε και είδαμε πόσο ε, δύσκολο είναι να αλλάξει η υιοθετημένη πράξη. Η απλούστευση αυτή πρέπει να γίνει με έχοντας λάβει υπόψη τη γενική αρχή όταν αριθμίζουμε τους ε, κανονισμούς για το 2000, μετά το 2030 και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα στους κανόνες αυτούς. Πριν τελειώσω να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το στόχο αυτών των τροπολογιών, ο οποίος μάλλον έχει χαθεί μέσα από τις διαδικαστικές αλλαγές και τις καθυστερήσεις στο Συμβούλιο του τελευταίους μήνες. Δεν είναι αυτό λάθος ούτε του Κοινοβουλίου ούτε της Επιτροπής μας να τονίσω. Ο αρχικός και τωρινό στόχος είναι να βοηθούν τα κράτη-μέλη και να υποφεληθούν από την πολιτική συνοχή σε μια κρίσιμη περίοδο και αν καθυστερήσει κι άλλο η έγκριση και η εισαγωγή των μέτρων για τις ε, επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, απλά θα έχουμε αργήσει. Οι αλλαγέ στη δεύτερη ανάγνωση θα ε, επιμηκύνουν πολύ περισσότερο αυτή τη διαδικασία και ίσως τελικά να εφαρμοστούν όλα αυτά αφού έχει φύγει η κρίση. Γι' αυτό ζητώ την υποστήριξή σας ε, σε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much indeed σα κατευχαριστώ κύριε Κυρίλοφ για την παρουσίασή σας. Τώρα θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτηση και δίνουμε καταρχήν το λόγο στην κυρία Ριάνταλ Κούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κύριλοφ για την επικοδομητική του εργασία. Επανειλημμένως είχα την ευκαιρία να σας αναφέρω την άποψη του ΕΛΚ Γι' αυτό μπορώ να είμαι τώρα σύντομη ως προς το τροποποίηση του κανονισμού 1083. Εδώ και μερικές μέρες άκουσα εκπροσώπους διαφόρων υπηρεσιών στην περιφέρειά μου που μου είπαν ότι θέλουν να εφαρμοστούν σύντομα τα μέτρα αυτά, παραδείγματος χάρη. Η αύξηση του κατοφλίου που προβλέπεται είναι πολύ καλή απλοποίηση και θα διευκολύνει όλα. Στα γαλλικά χρησιμοποιούμε μια έκφραση που λέει κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση του κύριου Κύριλοφ μάλλον παρά να αρχίσουμε μια συζήτηση που μπορεί να καταλήξει σε αδιέξοδο. Γι' αυτό δεν θα καταθέσουμε τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Ας εφαρμοστούν επιτέλους αυτά τα μέτρα απλοποίησης όσο το δυνατόν συντομότερα για τα, τις προβλεπόμενες πιστώσεις ήδη από το 7. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη μιλήτρια η κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό που τελικά έχουμε μία έκθεση. Έπρεπε να είχε γίνει και από πέρυσι. Τελικά τα καταφέραμε. Νομίζω ότι ο εισηγητής ουσιαστικά έχει ακολουθήσει το δρόμο του Συμβουλίου. Σε αυτή την έκθεση υπάρχουν κάποιες τροπολογίες τις οποίες γνωρίζει ήδη ο εισηγητής. Στις αρχές του Νοεμβρίου τις καταθέσαμε ε, ώστε να μπουν στην τελευταία τελική έκθεση. Δεν τις έχει υιοθετήσει εν μέρη και γι' αυτό θα καταθέσουμε αυτές τις τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο να είναι βιώσιμες οι επενδύσεις που γίνονται ε, να μην δίνει μόνο λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είναι και επιτυχημένα τα προγράμματα στις περιφέρειες, να είναι βιώσιμα η και ε, να καλύπτουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τους στόχους μιας βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που επιδιώκουμε κύριε Κυρίλοφ. Γνωρίζετε τις τροπολογίες εδώ και καιρό. Θεωρήσαμε ότι θα τις κάνατε θα τις υιοθετούσατε κι εσείς. Ε, εάν, ε, εφόσον λοιπόν δεν το κάνετε, θα θέσουμε αυτές τις τροπολογίες. Φίλε Ντάνκ, Φράου Σρέντερ, το λόγο έχει ο κύριος Αγκουράκης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα διαφωνήσω με τον εισηγητή και με τη γενική φιλοσοφία. Κατά τη γνώμη μου, ε, τα περιφερειακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοχής, κοινωνικά πέστε τα, κοινωνικά πέστε όπως θέλετε, όχι απλώς δεν αντιμετώπισαν την κρίση, κατά τη γνώμη μου την επιταχύναν κιόλα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αν θέλετε το κουβεντιάζουμε. Αυτό που ήθελα εγώ να σημειώσω τώρα στην ε, παρένθεση, στην σύντομη τοποθέτησή μου, είναι εξή. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχει μια τροπολογία του άρθρου 57, όπου γίνεται λόγος να αφαιρεθεί ε, μια διαδικασία χρηματοδότησης των επενδύσεων ή των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν. Ρωτάω, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Η εισήγηση είναι να φύγει η χρηματοδότηση των θέσεων εργασίας. Αυτό δηλαδή εισηγούμαστε. Και να μείνει μόνο να διατηρηθούν οι επενδύσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω καταλάβει εγώ καλά. Αλλά πάντως δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή κρίσης, σε μια εποχή έξαρσης της ε, ανεργίας και παρά το γεγονός, εγώ επιμένω ότι το Ταμείο Συνοχής και τα κοινοτικά περιφερειακά προγράμματα είναι πλήρως εναρμονισμένα και με την στρατηγική της Λισαβόνας και με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν είναι δυνατόν, λέω, σε συνθήκες τέτοιες, αν είναι έτσι, να αφαιρείται αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αγκουράκη. Νομίζω στο τέλος της συζήτησης ο, ο, κύριος Ραπορτέρ δώσει κάποιες ε, Uh, vreau sa mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Kirilov. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο εισηγητή Κύριλοφ ή μάλλον τον εισηγητή κύριο Κύριλοφ διότι και εμεί συμφωνούμε βασικά με τις τροπολογίες του γιατί βρίσκουμε ότι ανταποκρίνονται στις αποφάσεις της 20 Νοεμβρίου του Συμβουλίου. Νομίζω ότι ο κύριος Κύριλοφ δικαίως στο σχέδιο έκθεσής του αναφέρει τα δύο κύρια στοιχεία, απλοποίηση και αντιμετώπιση της κρίσης. Αν μιλήσουμε για την απλοποίηση, οι τροποποιήσεις που προτείνονται συμφωνούν απόλυτα με όσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή μας είχε προτείνει επανειλημμένως επαναλαμβάνω για την απλοποίηση των κανονισμών και γενικότερα την υπερβολική, υπερβολικά, τα υπερβολικά πολλά νομοσχέδια που επιβαρύνουν που εμποδίζουν μάλλον την πρόσβαση στα, σε τέτοιες χρηματοδοτήσεις. Τώρα για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης ο εισηγητής τροποποιεί την αρχική πρόταση της Κομισιόν για την προκαταβολή 2% του Ταμείου Συνοχής και άλλα 4% του Κοινωνικού Ταμείου και για μας αυτό είναι ικανοποιητική πρόταση. Συγχαίρομαι λοιπόν τον εισηγητή, θα τον υποστηρίξουμε ως φιλελεύθεροι και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να βοηθήσουμε πέντε κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πρόβλημα ήδη από τώρα, γιατί το χρειάζονται. Αν αρχίσουμε τώρα να αμφισβητούμε το μέλλον ή να συζητάμε καν το μέλλον της πολιτικής συνοχής, χάνουμε την κύρια ιδέα. Τώρα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι είχαμε πολλές ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε ακόμα να βελτιώσουμε και να κάνουμε πιο καλό το γενικό κανονισμό για τις περιφέρειες. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει αυτά να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας για τη συζήτηση, για τη μελλοντική συζήτηση για την ε, πολιτική συνοχής και να κάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι μπορούμε ε, γιατί εδώ έχουμε μία έκθεση η οποία θέλει να βελτιώσει την κατάσταση σε σχέση με την οικονομική κρίση με τις δυνατότητες που έχουμε. Λυπάμαι που η Κομισιόν και το Συμβούλιο πραγματικά χρειάστηκαν τόσο πολύ χρόνο και δαπάνησαν τόσο χρόνο για, και τράβηξαν πέρα από εδώ και από εκεί μια πρόταση που θα είχε τη δυνατότητα πλειοψηφίας εκ της αρχής και τελικά ο εισηγητής μας πήρε, αναγκάστηκε να κάνει αυτή την έκθεση τόσο αργά. Ελπίζω λοιπόν τώρα να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ώστε να εφαρμόσουμε τα μέτρα και να αντιμετωπίσουμε την κρίση και μετά ε, μπορούμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Είναι, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ευθύνη ε, να βοηθήσουμε τις περιφέρειες ε, και τα κράτη-μέλη να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να αποφασίσουμε και η συζήτηση για βασικά θέματα, όπως είπε και η συνάδελφος, μπορεί να ακολουθήσει λίγο αργότερα. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή που χρειάστηκε να συντονίσει τόσα πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και ε, συμφωνώ με την έκθεση, ελπίζω ότι θα ψηφιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Και εγώ ε, θα ήθελα να σας πω ότι ε, εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι ε, μπόρεσε να συντονίσει διάφορες προτάσεις ο εισηγητής και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η έκθεση η έκθεση ε, πραγματικά μιλά για ένα διαφανές και σαφές σύστημα ελέγχων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εις των δικαιούχων. Να προσθέσω όμως ότι Λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοπιστωτική κρίση που διανύουμε, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα έχουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και, να, και τα μέτρα κατά της κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν αρκετά χρήματα για περαιτέρω επενδύσεις στις περιφερειές τους. Είναι σημαντικό αυτό διότι πρέπει ε, να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόληση για τους πολίτες τους και τις επιχειρήσεις τους. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Κύριλοφ για κάποιες σύντομες παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου και εγώ να πω δύο λόγια στη μητρική μου, στα ελληνικά. Θα ήθελα και εγώ, κύριε Λόφ, να σας, να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε και να καλωσορίσω την έκθεσή σας. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως πολύ σωστά έθεσε ο εισογητής, έχουμε δύο επιλογές. Είτε να αποδεχθούμε την συμβιβαστική πρόταση που επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών μελών στις 30 Νοεμβρίου του 2009 και να προχωρήσουμε ώστε να μην χάσουμε και άλλο πολύτιμο χρόνο επιπλέον του εξαμήνου της ως τώρα καθυστέρησης, είτε να κάνουμε αλλαγές στην πρόταση, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω καθυστέρηση. Προσωπικά πιστεύω ότι στην σημερινή εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη λόγω της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή και να προχωρήσουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ώστε τα μέτρα αυτά να γίνουν πράξη το συντομότερο δυνατόν. At this point, I would like to give the floor to Mr. Kirillov. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις ε, ε, πολύτιμες παρατηρήσεις και για τη συμβολή σας. Είναι πολύ σημαντικό ε, για να δούμε κατά πόσον έχουμε την ε, αρκετό βαθμό υποστήριξη για να προχωρήσουμε ομαλά προς τα εμπρό. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες. Και βεβαίως χρειαζόμαστε αυτή την υποστήριξη αν θέλουμε, όπως σας είπα, να προχωρήσουμε προς τα εμπρό ομαλά. Βεβαίω, αν υπάρξουν τροπολογίε, ε, έχουμε την ε, συνηθισμένη διαδικασία και θα τι εξετάσουμε. Αυτό όμω το οποίο είναι σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι υπάρχει και τόσο βαθμό υποστήριξη για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ λοιπόν του σκιώδει εισηγητέ, την κυρία Κόβη, την κυρία Σρέντερ. Μία ερώτηση πρέπει να απαντήσω από τον, την ερώτηση του κυρίου Αγκουράκη που αφορά το άρθρο 57. Κοιτάξτε, θέλω να σας καθησυχάσω. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα το επικίνδυνο. Ασχολείται και αναφέρεται στους κανόνες που ε, αφορούν την παρακολούθηση ε, και ε, την ε, συνεχιζόμενη βάση. Και αυτό όλα υπολογίζεται από τη στιγμή που δημιουργείται η θέση απασχόλησης και όχι από τότε που θα κλείσει όλη η συνεργασία με βάση του υφιστάμενου άρθρου 57. Δεν, δεν αφαιρείται τίποτα. Και για άλλη μια φορά το όλο θέμα έχει να κάνει με την απλοποίηση των κανόνων. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλους για την πολύτιμη υποστήριξή σας, γιατί νομίζω ότι τη χρειάζονται όλες οι χώρες μας. Και όπως είπε η κυρία Βανέσκου, Ορισμένε χώρε χρειάζονται περισσότερο αυτή την υποστήριξη γιατί ε, βιώνουν μια ιδιαίτερα δραματική κατάσταση. Και βεβαίω ε, έχουμε τι πέντε χώρε που ανέφερα, τι ε, βαλτικέ δημοκρατίε, μάλλον την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, αλλά στο μεταξύ και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό σας λέω ότι ε, Ορισμένε χώρε επίγονται ιδιαίτερα, αλλά σε τελευταία ανάλυση όλε ε, οι χώρε ε, έχουν ανάγκη από τα μέτρα αυτά. Και νομίζω ότι θα είναι προ συμφέρον όλων εάν δράσουμε γρήγορα και καταλήξουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά για την παρουσίασή σας και σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση που έγινε. Πριν λοιπόν κλείσει η συζήτηση στο θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι σε αντίθεση με, τους, ε, με, τους, με τις άλλες νομοδοτήσεις της μερίσια διάταξη, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 25 Φεβρουαρίου σε 6 το απόγευμα, λόγω των χρονικών περιορισμών και το γεγονός ότι απαιτείται να διοργανώσουμε τριμερή διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επειδή λοιπόν ε, ε, ε, αυτό αφορά τη συγκεκριμένη κατάσταση. Το συγγνώμη, έχετε το λόγο. Κανονικό, οι σκιώδει εισηγητέ βρίσκονται και αυτοί στον τριμερή διάλογο κομμάτι τη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι σκιώδη εισηγήτρια και δεν ξέρω ημερομηνίε ή πληροφορίε για τον τριμερή διάλογο. Ίσως ο εισηγητή να μα δώσει κάποιε πληροφορίε τώρα. Yeah. Mr. Kirillov. Κύριε Κύριλο, κοιτάξτε. Είχαμε μία άτυπη συνεδρίαση μέχρι στιγμής, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει με τις τροπολογίες. Είναι αλήθεια ότι η κυρία Σιραντέρ πριν από λίγο καιρό μου έστειλε τις προτάσεις της, αλλά ε, ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ακολουθούμε τη διαδικασία όπως πρέπει. Πάντως, ε, Ελπίζω όλοι να καταλάβουμε ότι μάλλον θα πρέπει να αποφύγουμε παράταση, δεύτερη ανάγνωση κτλ. Ευχαριστώ κύριος Βανίστεροι. Ευχαριστώ. Μέχρι στιγμή πραγματικά πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα στην ολοκλήρωση αυτού του θέματο και όχι τώρα το κάνουμε πιο περίπλοκο. Σα παρακαλώ. Οπότε, εγώ θέλω να μου πείτε το εξή. Σε ποια ολομέλεια ε, να στρέψουμε την προσοχή μα. Και θέλω να ασκήσω πίεση και στο, να ασκήσουμε πίεση και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ε, προ την κατεύθυνση αυτή. Εγώ δεν άκουσα κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ψηφίσουμε. Ήδη έχει γίνει αναβολή. I'm just informed that the plenary από ό,τι ενημερώνομαι, η, η, η σχετική ολομέλεια θα είναι η ολομέλεια του Απριλίου. I'm Σε ζητώ συγγνώμη. Κοιτάξτε, εάν έχουμε μία ανάγνωση, ο τρίλογος γίνεται στο χρονικό διάστημα μετά την Επιτροπή, μετά τι ψηφοφορία στην Επιτροπή και μέχρι τα λομέλια Ακούσαμε τον, τον τρίλογο, τον τριμερή διάλογο και εγώ δεν έχω λάβει καμία πληροφορία. Okay. We will uh, inform you later. Ωραία, θα σε ενημερώσουμε αργότερα. Let's move. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, απαλλαγή 2008. Γενικός Προπολογισμό, τμήμα 3, Επιτροπή. να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιάν Όλμπιχτη που είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο. Ε, ε, Χρησιμοποιήσω τη μητρική μου. Ε, właśnie trwają prace w Komisji Kontroli Budżetowej dotyczące Εργαζόμαστε στην Επιτροπή, ε, οι εργασίες στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου συνεχίζονται για την απαλλαγή 2008 ε, στο τμήμα 3, την Κομισιόν και τις εκτελεστικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία μιας γνωμοδότησης η οποία θα δοθεί στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Είμαστε υπεύθυνοι ε, να προτείνουμε Ε, κάποιες ε, κατευθύνσεις ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό το κείμενο για το οποίο συζητάμε σήμερα αναφέρεται σε διάφορα κείμενα πηγές στα οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Πρώτον, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου η οποία ε, εκδόθηκε, δημοσιεύθηκε στην ε, επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευχός ε, C269. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αναλύεται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Το δεύτερο σημαντικό έγγραφο στο κείμενο που προτείνω αναφέρεται ως κάτι το οποίο αδειμονούμε να λάβουμε. Θα το βρείτε στο σημείο 2 των προτάσεών μου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι έχει δημοσιευθεί ήδη το έγγραφο. Πρόκειται για το έγγραφο της 18ης Φεβρουαρίου και ο τίτλος είναι οι επιπτώσεις του σχεδίου δράσης ε, στην ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Κομισιόν και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευθεί για να καταδείξει τις επιπτώσεις του σχεδίου δράσης στο σχέδιο δράσης που αναφέρεται σε όλα τα άλλα έγγραφα. Εδώ βλέπουμε πληροφορίες σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής του Διαρθρωτικού Ταμείου ως αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει αναφερθεί στις βελτιώσεις αυτές και στο σχέδιο δράσης και στο παρελθόν. Ως συντάκτης της γνωμοδότησης θα κάνω ο ίδιος μια τροπολογία. Θα αλλάξω το σημείο 2, διότι δεν μπορούμε πλέον να δημονούμε για να λάβουμε, να λάβουμε τη δημοσίευση. Ε, αναφέρομαι ξεκάθαρα λοιπόν στο κείμενο, στο κείμενό μου στο έγγραφο και δίνονται οι πληροφορίες ε, που λένε ότι ως αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο της Επιτροπής αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την ίδια διαδικασία όπως και το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρει ότι το επίπεδο λαθών μειώνεται από το 11% στο 5% και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Γι' αυτό και καταθέτω αυτή την τροπολογία. Και λέω ότι η Επιτροπή μας καλωσορίζει το γεγονός πως μπορούμε πλέον να παρατηρήσουμε τα θετικά αποτελέσματα του σχεδίου δράσης. Το έγγραφο είναι εντελώς καινούριο. Μόλις το έλαβα. Γι' αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμη η τροπολογία μου. Θα την κάνω όμως. Στην γνωμοδότηση να πω ότι από τη μία λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που ε, δίνονται από το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με κάποια ασφάλματα στα προγράμματα, στο project από την άλλη, στην γνωμοδότησή μας προτείνουμε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να ελέγξει συγκεκριμένα τους λόγους που εμφανίζονται αυτά τα σφάλματα. Ειδικότερα θέλουμε να δώσουμε έμφαση στα σφάλματα που γίνονται στις διαδικασίες δημοσίων προεμιθειών. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια συζήτηση που λαμβάνει χώρα ε, αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα και ο Σάλφος Βλάζακ επίσης ε, ετοιμάζει μία γνωμοδότηση για αυτό το θέμα. Να τονίσω επίσης ότι η πολιτική συνοχής χρησιμοποιεί ε, ιδιαίτερα μέσα, χρηματοδοτικά μέσα για τη διαχείριση που ναι μεν δίνουν πολλές ευκαιρίες, απ' την άλλη όμως γύρουν και πολλές δυσκολίες. Η γνωμοδότηση επίσης προτείνει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των σφαλμάτων και των καταχρήσεων που ε, πρέπει να αναλύονται και μετά να υπόκεινται σε ειδικέ διαδικασίες, ειδικότερα στα πλαίσια της Όλαφ. Γι' αυτό και στο σχέδιο που έχω συντάξει. ευχαριστώ την προσοχή σας καταρχάς από τη μία σε επικριτικές παρατηρήσεις, αλλά από την άλλη και σε θετικά σχόλια. Να επιστήσω την προσοχή σας στη βελτίωση. Η βελτίωση είναι ξεκάθαρη υπό το φως του νέου γράφου. Επίσης η αλλαγή στις τάσεις η τάση για τη μείωση του επίπεδου των σφαλμάτων και την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων. Η γνωμοδότησή μας λοιπόν που θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και σχετίζεται με το τμήμα 3 Πολιτική Συνοχής και Διαρθρωτικά Ταμεία αν η Επιτροπή μας αποδεχθεί τις παρατηρήσεις μου θα προσπαθήσουμε να πείσουμε την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να τις κάνουν αποδεκτές και να τις συμπεριλάβουν στο εγγραφό του. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ισηγητά για την παρουσίασή σας. Τώρα θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτηση και πρώτος το λόγο έχει ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Θα ήθελα να ε, σημειώσω ευθύ εξ αρχή ότι το οικονομικό έτος του 2008 δεν παρουσίασε βελτίωση σε σύγκριση με το 2007. Επίσης ε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον ένα 11% του προϋπολογισμού του συνολικού ποσού του ε, Ταμείου Συνοχής που καταβλήθηκε το 2008 δεν θα έπρεπε να έχει καταβληθεί. Αυτό το σχολιάσαμε και άλλη φορά. Ε, φαίνεται όμως πως πρέπει να γίνει ξανά αναφορά ότι η παραπέρα μείωση των ε, ρυθμών σφαλμάτων εξακολουθεί ή θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Βέβαια μιλούμε κομψά για ε, λάθη, για σφάλματα. Είχαμε μιλήσει και για τρεις χώρες, οι οποίες δεν κατονομάστηκαν και όπως ε, επισημαίνεται και στο σημείο 7 από τον συντάκτη της γνωμοδότησης ε, δεν κοινοποιήθηκε κανένα κρούσμα απάτης και έτσι όταν μιλάμε για σφάλματα ε, δεν παραπέμπουμε κατανάκιν σε αυτήν. Θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο το πράγμα, ε, ιδιαίτερα όταν ζούμε σε μια περίοδο όπου εγκαλούνται χώρες για σφάλματα ή αποκαλύπτεται με αφορμή την περίπτωση της Ελλάδας ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παραπλήσεις τακτικές είναι λυπηρό λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το γεγονός ότι η επιτροπή προτίθεται να περιμένει ως το 2012 πριν υποβάλει πρόταση αναφορικά με τον ανεκτό κίνδυνο σφαλμάτων στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι καθώς η προγραμματική περίοδος 2000-2006 πλησιάζει στο τέλος της, τα κράτη-μέλη με την πίεση να απορροφήσουν το σύνολο των ε, δεσμευμένων κονδυλίων μπορεί να έχουν υποβάλει έναν ε, αυξημένο αριθμό απρόβλεπτων έργων. Επίσης, το ελεκτικό συνέδριο διαπιστώνει την ε, αργή εκκίνηση των προγραμμάτων που σχετίζονται με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 λόγω της καθυστερημένης υποβολής εκ μέρου των κρατών μελών των εκθέσεων αξιολόγηση συμμόρφωσης και των στρατηγικών ελέγχων. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τα συστήματα ελέγχου να αποτύχουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό των σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας φάσης. Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή, ας το πούμε έτσι, κατονομάζω και διαπέμπω, διαπομπεύω. Αυτό είναι μία άμυνα. Στις ε, εκθέσεις τους θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τα κράτη-μέλη, τα συστήματα ελέγχου, των οποίων είναι τα λιγότερο αποτελεσματικά. Και είπαμε, η περίοδος αυτή προσφέρεται πάρα πολύ για να γίνει κάτι τέτοιο. Και αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες το σύστημα των δημοσιονομικών διορθώσεων πρέπει να γίνει πιο αποτρεπτικό. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, κάθε μη επιλέξιμη δαπάνη που προσδιορίζεται από την Επιτροπή ή το Ελεκτικό Συνέδριο μπορούν να αντικατασταθούν αμοιβαία με επιλέξιμες δαπάνες από ένα κράτος μέλος. Θα πρέπει να εξετάσουμε ένα σύστημα με το οποίο στο μέλλον μόνο παρατυπίες που εντοπίστηκαν από τα ίδια τα κράτη-μέλη και όχι από άλλον, να μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες δαπάνες όπου δεν θα υπάρχει απώλεια της χρηματοδότησης για τον λόγο κράτος μέλος. Είναι και αυτό μια τακτική άμυνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ε, να τονίσω ότι ο Γιάνν Όλμπρεχτ, ο εισηγητής, μας έδωσε μια ιδέα για το τι συμβαίνει, ποια είναι τα λάθη που έχουν γίνει και για τις βελτιώσεις που έχουν προταθεί και εισαχθεί να υπογραμμίσω το γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος για να εξετάσουμε αυτό το νέο έγγραφο. Ζητήσαμε αυτό το σχέδιο δράσης στην περασμένη νομοθετική περίοδο και γι' αυτό θέλω να βεβαιωθώ ότι αυτό θα αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Οι βελτιώσεις που αναφέρονται στην τρέχουσα περίοδο, ε, όπως και στο 2008, είναι αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την προηγούμενη περίοδο. Ζητώ να εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες που έχουμε και τις πληροφορίες που έχουμε λάβει ο σημείωση για να μπορέσουμε η γνωμοδότηση που θα δώσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να οδηγήσει στο να έχουμε πιο θετικές τάσεις από αυτές που βλέπουμε ήδη στα νούμερα. Ο κύριος Όλμπριχτ θεωρώ ότι έχει φτιάξει μία ε, καλή έκθεση και μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μανέσκου. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ε, ευχαριστούμε τον κύριο Όλμπριχτ για το έγγραφο το οποίο μας παρουσίασε. Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη η άποψή του και, λεπτομερό, και εκτίθεται λεπτομερός και δείχνει τις ελλείψεις που χαρακτήρισαν το χρονικό 2000-2006 όσον αφορά τις πληρωμές. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το 2008 δείχνει ότι οι ενδιάμεσες πληρωμές καθώς και τα επιχειρησιακά προγράμματα παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση ενώ η έκθεση για το 2000-2006 χαρακτηρίζεται από υψηλό αριθμό σφαλμάτων όσον αφορά τι πληρωμέ που πραγματοποιήθηκαν. Λοιπόν, για όλου αυτού του λόγου πιστεύουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο θα έπρεπε να δώσει έμφαση στον έλεγχο της αποδοτικότητας των ε, προγραμμάτων. Δεν αρκεί η ανάλυση συμφωνίας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, περαιτέρω και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των ταμείων. Τα διευθυντικά ταμεία και ε, το Ταμείο Συνοχή και οι πληρωμέ που γίνονται στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνε με του κοινοτικού κανόνε, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται ε, ε, στο βασικό, στους βασικούς στόχους των κρατών μελών και στους στόχους των ίδιων των, προγραμμάτων. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο εν λόγω δημοσιονομικός κανονισμός που αφορά τη χρηστή ε, δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει να μας, ε, ε, να μας οδηγήσει στο δρόμο της εξέτασης της ε, οικονομικής αποδοτικότητας, δηλαδή να ελέγξουμε κατά πόσον τα συγκεκριμένα κονδύλια δαπανήθηκαν όπως έπρεπε και κατά πόσον επετέφθηκαν οι στόχοι των προγραμμάτων. Είναι απλό. Νομίζω ότι η άποψη του κύριου Όλμπριχτ είναι απόλυτα ορθή δεδομένων όλων αυτών των στοιχείων. Και θα τον υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ja, Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την έκθεση του κ. Όλμπριχτ, πρέπει να πούμε ότι είναι καλή. καλή. Και αναγνωρίζουμε επιτέλους την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Δηλαδή ότι τώρα τα σφάλματα είναι λιγότερα ενώ ταυτόχρονα έχουμε και καλύτερα μέσα. Αλλά επιτρέψτε μου να εκφράσω ορισμένες ε, ανησυχίες, γιατί πάντα τα ίδια κράτη-μέλη είναι αυτά που φαίνεται ότι διαπράττουν τα ίδια σφάλματα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο ε, ανταμοιβή των κρατών μελών ε, που για πολλά χρόνια δεν διέπραταν αυτά τα σφάλματα και ίσως δεν θα έπρεπε να ελέγχονται πλέον ενώ άλλα κράτη-μέλη τα οποία επανειλημμένα ε, έχουν διαπράξει σφάλματα συμμόρφωσης ίσως θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτική βάση. Γιατί λοιπόν στην Επιτροπή τώρα, τώρα γιατί στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν ε, λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με, ε, ε, με ένα μέσο το οποίο αναπτύσσεται και με την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που αναφέρει ότι τα χρήματα αυτά δεν δαπανήθηκαν όπως θα έπρεπε. Εμείς λοιπόν ως Επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης θα έπρεπε να λέμε περισσότερο τη γνώμη μας αν θέλετε για το πώς πρέπει να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίπερ. Όπως θα καταλάβατε το θέμα ο φάκελος έχει διανεμηθεί λοιπόν. Όμπερ Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η... Το σχέδιο έκθεσης δείχνει ένα ποσοστό των λαθών που γίνονται, ειδικότερα όσον αφορά τις ε, καταβληθήσεις ε, πληρωμές. Ε, νομίζω ότι ε, υπάρχουν πολλά λάθη τα οποία δεν έχουν να κάνουν με απάτη αλλά γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Σε όλη τη συζήτηση πρέπει να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι την εποπτεία την έχει η Κομισιόν. Όμως και τα κρατημέλη έχουν σημαντική ευθύνη για τον έλεγχο συγκεκριμένων εργασιών. Είναι λοιπόν σημαντικό τα διάφορα επίπεδα ελέγχου να δρουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε πολύ περίπλοκες ρυθμιστικές διατάξεις, νομοθετικές διατάξεις και πολλές φορές ε, γίνονται σφάλματα ε, χωρίς να είναι σκεμμένα. Και γι' αυτό ε, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας και να σκεφτούμε ε, εάν ε, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα εκπαίδευσης μέχρι και στο τελευταίο κρίκο αυτής της αλυσίδας ε, ώστε να αντιμετωπίζονται τα διάφορα επίπεδα. Επίσης υπάρχει και ένα σύστημα μπόνους για αυτούς που δεν κάνουν σφάλματα και αυτό θα ήταν καλό σε, σε αυτούς τους κανονισμούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Ομπερ Πριν... Λοιπόν, ε, έχουμε τον κύριο Σωμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πριν δώσουμε το λόγο, θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Και θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τη, γνωμάτευση, τη γνωμοδότηση συγγνώμη, του κυρίου Όλμπριθ και να τον συγχαρώ για τη δουλειά του. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση που αντικατοπτρίζει με ρεαλιστικό τρόπο, θα έλεγα, την πραγματικότητα και περιέχει όλα τα κρίσιμα σημεία και πτυχές που καθορίζουν ή δύναται να καθορίσουν το ποσοστό λάθους, κάνοντας ταυτόχρονα όλες τις απαραίτητες επισημάσεις στις οποίες θα πρέπει να βασιστεί η δινεται να καθορισουν το ποσοστο λαθους κανοντας ταυτοχρονα ερμηνεία αξιολόγηση των ποσοστών που καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω στην εξαιρετική γνωμοδότηση του κυρίου Όλμπριχτ είναι στο σημείο 4, όπου θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο της απλοποίησης στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων ως καθοριστικού παράγοντα για την περαιτέρω μείωση του ποσοστού λάθους. Μιας και όπως είναι γνωστό σε όλους μας και όπως αναφέρεται άλλωστε και στην γνωμοδότηση, δεν είναι εύκολο για όλους τους φορείς να ανταποκριθούν στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις αν δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ικανότητα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, αν και ήδη αναφέρεται ξεκάθαρα στην γνωμοδότηση. Πρέπει πάντα... Okay. I'm sorry for that. Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για λάθη και όχι για απάτη, γιατί στις συζητήσεις που κάνουμε στο πλαίσιο της ΚΟΝΤ για την απαλλαγή του 2008, ορισμένοι συνάδελφοι συχνά συγχαίουν το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο, άρα κύριε Όλμπιρ θα εκθέσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ε, να το συντομία στις διάφορες παρατηρήσεις των μελών τη επιτροπή μα. Πρώτα απ' όλα, και εγώ είμαι μέλο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και ε, ελέγχου του προπολογισμού. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το τι ελέγχουμε στην ουσία. Αυτά που είπε και η κυρία Μανέσκου. Ελέγχουμε τις διαδικασίες. Το κατά πόσον τα πάντα είναι εντάξει ως προς τα δεδομένα, τα έγγραφα ή Την αποτελεσματικότητα. Και βεβαίως ε, αυτή είναι η έκθεση ε, ελέγχου του προπολογισμού. Άρα στην ουσία αφορά τι διαδικασίε και όχι την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα. Η συνεχιζόμενη συζήτηση με το ελεκτικό συνέδριο είναι το πώ μπορούμε να υπερπηδήσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να μην συζητάμε μόνο τι διαδικασίε αλλά και την αποδοτικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν υπάρχει σαφή απάντηση σήμερα. Το, ε, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Δεν ήθελα να το πω σε αυτή τη γνωμοδότηση δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρξε απάτη, διότι και βεβαίω και υπάρχει. Αλλά σε αυτό το περίφημο 11% αυτά τα παραδείγματα δεν παρουσιάστηκαν ως απάτες, αλλά ως λάθη. Οπότε, αυτά τα οποία βλέπουμε στα έγγραφα της Επιτροπής είναι ότι Όσον αφορά αυτόν τον αριθμό των λαθών, δεν έχουν στοιχεία για απάτε. σω υπάρχουν κάπου αλλού, αλλά δεν, ε, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ποσοστό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ιδιαιτερότητα τη πολιτική συνοχή είναι το εξή. Υπάρχουν τα έργα, τα σχέδια και μετά οι πληρωμές που γίνονται από τα κράτη-μέλη από τι εθνικέ αρχέ που κάνουν τι πληρωμές, στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχο, τα λάθη και φυσικά οι διορθώσεις. Και στο τέλος του έτου ή μετά από τη συνολική περίοδο. Άρα λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο παίρνει για παράδειγμα, εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση, τη χρονική στιγμή χ, ελέγχουν και βλέπουν αυτό το 11% για παράδειγμα. Όμω εδώ έχουμε πολυετή προγραμματισμό και βεβαίω υπάρχουν και οι δημοσιονομικέ διορθώσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το πούμε ότι ένα, το πρόγραμμα δράσης το οποίο εισήχθη δείχνει τώρα δείχνει ότι ε, οι δημοσιονομικές διορθώσεις γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Πρέπει να πω ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις που είχαν ήδη γίνει από την Επιτροπή είναι μεγαλύτερες από ό,τι στο χρονικό διάστημα 2000-2006. Θέλω να πω δηλαδή, ε, πέρυσι ήταν περισσότερες οι διορθώσεις από ό,τι προηγουμένως. Και καταλαβαίνετε τι προσπάθεια κατεβλήθηκε. Κάτι άλλο το είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας είναι το εξή. Όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες, Στην τελευταία ανάλυση ποιος είναι ένοχος. Έχουμε κακό ή κακό ε, σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες ή το σύστημα είναι καλό και η υλοποίηση είναι κακή. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τι κρατικέ προμήθειε. Άρα το ερώτημα είναι τι συμβαίνει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα τη ε, πολιτική συνοχή. Γι' αυτό η Επιτροπή μα πρέπει να δείξει ότι όλα τα λάθη δεν είναι συστηματικά λάθη τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην πολιτική συνοχή, αλλά συνδέονται με την πολιτική συνοχή. Δηλαδή ότι δεν φταίει η πολιτική συνοχή σε αυτή καθεαυτή αλλά η διαχείριση. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη δεδομένου ότι αυτή η πολιτική είναι απολύτως αναγκαία. Αυτό ήθελα και εγώ να αποδείξω αυτή την πολύ σύντομη γνωμοδότηση και να σας δείξω ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε τα λάθη βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε τις αλλαγές, τις θετικές αλλαγές και να ζητήσουμε από την Επιτροπή για παράδειγμα το εξή. Καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει το γιατί ε, οι κρατικές προμήθειες αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλα τα κρατημέλη. Οι διορθώσει μπορεί να αφορούν κυρίω ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά βεβαίω αυτό δεν είναι το θέμα και το αντικείμενο τη συγκεκριμένη έκθεση. Ακριβώ για αυτό το λόγο, από πολιτική άποψη, εγώ συντάκτη γνωμοδότηση βεβαίω, πρέπει ε, πιστεύω ότι πρέπει εμεί ω Επιτροπή να δείξουμε, ε, ω Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, να δείξουμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα σε κάθε διαδικασία, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν συνδέονται με την πολιτική συνοχή σε αυτή καθε αυτή. Συνδέονται με τι διάφορε διαδικασίε. Γι' αυτό αυτή η έκθεση δείχνει και την καλή όψη και την κακή όψη. Okay, thank you very much indeed, Mr. Σας κατευχαριστούμε κύριε Ισηγητά καθώς και όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Επειδή όμως δεν χρειάζεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, προχωράμε στο επόμενο σημείο το 6. Δηλαδή έκθεση από τις ανακοινώσεις της Επιτροπής κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών κατασυτοροφών. Ε, μάλιστα κύριε Όλμπριχτ, συγγνώμη αλλά δεν το λέει εδώ το χαρτί μου. 1η Μαρτίου λοιπόν, εντάξει, να το γράψω. 1η Μαρτίου, το καταλάβατε όλοι και όλες, μάλιστα. Είπαμε τώρα το 6 έκθεση της ανακοινώσεως της Επιτροπής Κοινοτική Προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Εισηγητής ο κύριος Βίκτορ Ουσπάσκης, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω λιθουανικά. Το θέμα το αναλύσαμε με εμπειρογνώμονες όπως γνωρίζετε και η αρμόδια επιτροπή επί είναι η Επιτροπή Περίβ, ΕΝΒΗ. Από την ανάλυση λοιπόν αυτή θα κάνουμε και εμείς τη γνωμοδότησή μας με αυτή τη βάση δηλαδή και θα σας αναλύσω με τη σειρά μου ορισμένες πτυχές που νομίζω ότι πρέπει να αναφέρονται στην γνωμοδότηση αυτή για την έγκριση της κοινή κοινοβουλευτικής θέσης για την πρόληψη των ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών. Θέλουμε να αυξηθεί ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων και Είμαστε πεπισμένοι ότι ένας ενεργότερος ρόλος των αρχών αυτών είναι απαραίτητος και για τον καθορισμό και την πρόληψη που είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης ώστε να εφαρμοστούν οι πιο απλές και λειτουργικές και αποτελεσματικές λύσεις. Επίσης, είναι σημαντικός ο ρόλος της διαβούλευσης και με δημόσιους και με ιδιωτικούς παράγοντας Βέβαια, οι επιπτώσεις των καταστροφών δεν περιορίζονται, δεν μειώνονται στα σύνορα κάποιου κράτους ή μιας περιφέρειας, αλλά η ταύτιση των κινδύνων για τέτοιες καταστροφές με βάση συγκεκριμένες περιφέρειες μπορεί να αποτελέσει τη βάση της πρόληψης. Φυσικά δεχόμαστε την πρωτοβουλία της Κομισιόν για καλύτερη και περισσότερη πρόληψη και συμπερίληψη τέτοιων προγραμμάτων στα μελλοντικά μας προγράμματα. Πρέπει μέχρι το 2013. Η χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων να αποτελέσει τον μοχλό ώστε να μπορούν τέτοια προγράμματα αντιμετώπισης να εφαρμόζονται σύντομα χωρίς καθυστερήσεις. Ε, βέβαια χρειάζεται και συντονισμός, αυτό είναι προφανές. Επίσης προτείνω να υποστηρίξουμε την ιδέα η χρηματοδότηση έργων υποδομών από τα διαρθωτικά ταμεία στις επόμενες προγραμματικές περιόδους να γίνεται με τον όρο να εφαρμόζονται πράγματι συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης. Αυτά σύντομα. Βέβαια η γνωμοδότησή μου έχει σταλεί σε όλους και μπορείτε να τη δείτε άμα θέλετε και γραπτός. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τρεμόπουλο. Συζητούμε για ένα θέμα κύριε Πρόεδρε το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα εφόσον ε, ζούμε ήδη τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Συμφωνούμε με το σχέδιο γνωμοδότησης γύρω από το ζωτικό ρόλο που έχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαχείριση των ε, φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τη σημασία των συντονισμένων ενεργειών μεταξύ των διαφόρων κλάδων και περιφερειών. Βέβαια, οι περιφέρειες δεν είναι το ίδιο ευάλωτες. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχει η διάσταση της συνοχής στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αναγκαία η αναθεώρηση των κανονισμών του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα πιστεύουμε πως αυτό πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία, να αξιοποιηθεί για την αποκατάσταση των ε, περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο και να ενσωματωθεί σε αυτό η παράμετρος της πρόληψης. Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική που θα περιλαμβάνει την αποτροπή των κινδύνων. Θα λέγαμε στα ελληνικά να είμαστε περισσότερο προμηθείς παρά επιμηθείς. Τώρα δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις λοιπόν και στην εποχή των κλιματικών αλλαγών ε, θα έχουμε ολοένα και περισσότερο έντονα ε, φυσικές ε, καταστροφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανώσει την ετοιμότητά της μέσα από την εφαρμογή των εργαλείων πρόληψης και αποτροπής σε τομείς ιδιαίτερα όπως η γεωργία και η δασοπονία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την ετοιμότητα πολιτικής προστασίας των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, τις ε, ακούσαμε επανειλημμένα και σε, ε, άλλες ε, διεργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως χρειάζονται αναβάθμιση. Χρειαζόμαστε επίσης νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση μιας ουσιαστικής ευρωπαϊκής δύναμης ανταπόκρισης στις καταστροφές. Και ιδιαίτερα, εφόσον ε, το είδαμε και το καλοκαίρι που πέρασε, για τα δασικά οικοσυστήματα της Νότιας Ευρώπης χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασία τους που θα εξασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση των μέτρων πρόληψης, αποκατάσταση, ναι, αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και προσαρμογή δυστυχώς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόπουλε. The next speaker is... Ο ε, επόμενος μιλητής, ο Λόπε. Thank you. Uh, no. Η dauguma dabar išsakytų pasiūlymų arba aspektų. The ε, Με συγχωρείτε. Τον κύριο Λοπέ Φοντανιά, ε, την κυρία Λοπέ Φοντανιά είπα εγώ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή όσον αφορά το ρόλο που αναπτύσσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Διότι ε, οι αρχές αυτές είναι αυτές που παρεμβαίνουν σε πρώτο επίπεδο για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταστροφών. Αλλά κοιτάξτε, οι καταστροφές, ε, το φαινόμενο των καταστροφών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο από την περιφερειακή διάσταση, ούτε καν από την εθνική. Ε, το φαινόμενο αυτό απαιτεί μια αποτελεσματική απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να ολοκληρώνονται και να ενισχύονται οι δράσεις των εθνικών ή των περιφερειακών αρχών και των τοπικών. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδε να ε, υπάρξει ένα πρωτόκολλο, ενιαίο πρωτόκολλο δράση για κάθε είδο καταστροφή, έτσι ώστε να υπάρξει η εγγύηση απόλυτη αλληλεγγύη ανάμεσα στι χώρε μέλη για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα να υποστηριχθούν ιδιαίτερα οι περιφέρειε με διαρθρωτικέ δυσκολίε, που είναι πολύ περισσότερο ευάλωτε απέναντι σε τέτοιου είδου φαινόμενα, διότι έχουν λιγότερου πόρου και μέσα για να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα αυτά. Επίση, θα πρέπει, ε, όπω άλλωστε είπε και ο ίδιο ηγητή, να δράσουμε στο επίπεδο πρόληψη και κυρίω στη βελτίωση του συντονισμού των διαφόρων ε, εμπλεκομένων που ε, παρεμβαίνουν στην πρόληψη και διαχείριση των καταστροφών. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα πρωτόκολλο συντονισμού των διαφόρων μέσων και των διαφόρων ε, ταμείων και κονδυλίων. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις ε, με την συνδρομή των νέων τεχνολογιών. Άλλο σημείο. Πρέπει να ξαναδούμε τα ε, δημοσιονομικά κονδύλια τα οποία ε, αφορούν, ε, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόληψη αυτών των καταστροφών. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την κατανομή των κονδύλιων αυτών έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του. Και τέλο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασία των δασών. Με δύο προτάσει οδηγία για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και για την, την, να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της ξηρασίας, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός των πολιτικών των κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα και να βελτιστοποιηθούν τα κοινωνικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Τέλο, επίση, θα ήταν ε, χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την ξηρασία και την απερίμωση, ε, για τι πλημμύρε ε, και για τι υπόλοιπε επιπτώσει των κλιματολογικών μεταβολών, έτσι ώστε να συλλέγονται πληροφορίε και να υπάρξει σωστή πρόληψη. Και προ αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσω και εγώ να συμβάλλω με τι παρατηρήσει Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να σας ζητήσω αν θέλετε να είστε σύντομοι για να είμαστε και μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βλάσακ. Eh, ε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, με εκπλήσει το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στρατηγικό υλικό για να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα και γι' αυτό καλωσορίζω αυτό το έγγραφο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά φυσικά δεν ασχολείται με την πρόληψη ή τις βέλτιστες πρακτικές και ένα σύστημα προειδοποίησης. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασυνδέσουμε τα μεμονωμένα project, ειδικότερα στις συνοριακές περιοχές αυτά πρέπει να διασυνδέονται και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται γιατί οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες κτλ. είναι φυσικές καταστροφές χωρίς σύνορα. Και εδώ να τονίσω και το θέμα της διεθνής αρρωγής. Θα πρέπει να υπάρχει ε, συντονισμός και έλεγχος αυτής της αρρωγής. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πίπερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για αυτή την θέση που πραγματικά δίνει μια άποψη για τις ε, ε, δίνει την άποψη των περιφερειών, εφόσον είμαστε Επιτροπή Περιφερειών και αυτό είναι ειδικότερα καλό γιατί ε, σχετίζεται με το τι συμβαίνει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Για τις τροπολογίες που αναφέρονται, δεν αναφέρεται γιατί χρειάζεται ε, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να σταματήσουμε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον υπάρχουν άλλα κίνδυνα τα οποία πραγματικά με τα οποία δεν μπορώ να ε, συνταχθώ. Γιατί χρειαζόμαστε χρήματα για την πρόληψη. Αυτά μπορούμε να τα ε, βρούμε στο πρόγραμμα της ε, περιφερειακής ανάπτυξης όταν οι χώρες χρησιμοποιούν τα χρήματα που έχουν για την πρόληψη μέσα από αυτό. Παρακαλώ, αφήστε τα επιχειρήματα όπως έχουν από την άποψη των περιφερειών. Επίσης, αν πέσει ε, ένα παιδί στο νερό ε, και πρέπει να κάνουμε κάτι, ε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Όταν έχουμε όμω ε, αεροπλάνα, πλοία κτλ. πρέπει να συντονίσουμε. Χρειαζόμαστε σχέδια, αλλά όχι νέους νόμους. Χρειαζόμαστε βέλτιστες πρακτικές. Γιατί η πάταξη των, πυρκαγιών, των δασικών πυρκαγιών είναι καλύτερη σε κάποιες χώρες από τις σε άλλες. Ίσως χρειαζόμαστε καλύτερη εκπαίδευση, όχι όμως νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και γι' αυτό θα, μείνω με την, θα συνταχθώ με τη γραμμή σας. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ κύριε Σόμπερμαϊερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είμαι σύντομος. Η, η ανάλυση είναι σωστή και η αλληλεγγύη σωστή επίσης. Είναι σημαντικό ότι ε, όταν υπάρχουν πυρκαγιές, όταν υπάρχουν πραγματικές καταστροφές, ε, υπάρχουν δυνατότητες ε, περιορισμού μέσα από τα μέσα που διατίθονται. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η διαχείριση καταστροφών να εμπλέκει και τους εθελοντές ε, οι, οποίες, ε, οι οποίοι μπορούν ε, και σε διεθνές επίπεδο να δράσουν και Νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, σε επίπεδο πρόληψης, αν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα σε σχέση με την χρήση εθελοντών για την πρόληψη καταστροφών στις περιφέρειες. Έτσι λοιπόν εδώ θα ήταν χρήσιμη η ανταλλαγή πληροφοριών και των ε, κοντιλίων που έχουν στη διάθεσή τους ε, οι χώρες. Επίσης σημαντικό είναι να πάρουμε μαθήματα από το παρελθόν. Ειδικότερα για συστήματα έγκαιρης ε, προειδοποίησης θα ήταν καλή η συνεργασία, όπως επίσης και σε επίπεδο έρευνας. Όμως αυτό πρέπει να το προωθήσουμε περαιτέρω. Επίσης, σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ο οποίος ε, θα πρέπει και αυτός να εμπλέκεται στην ε, πρόληψη, να εκπαιδεύεται εγκαίρος. Στην ε, Αυστρία, για παράδειγμα, έχουμε τέτοια εκπαίδευση ήδη από το σχολείο για τις ε, φυσικές καταστροφές, ε, ειδικότερα στο Τυρόλο. Παιδιά στο σχολείο μπορούν ε, από πολύ μικρά να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τόγερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να υποστηρίξω την προσέγγιση του, του εισηγητή ότι θέλουμε μία ε, περιφερειακή προσέγγιση και να είμαστε συνεπείς σε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή ότι ε, μπορεί να γίνει επιτόπου να μην γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήταν λάθος η συζήτηση αν πηγαίναμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα, η οποία έκανε τόσες ε, παραβάσεις, προβλήματα με τις στατιστικές. Τώρα έχουμε αιτιάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η οποία δεν έλεγξε την κατάσταση. Τώρα και για τις πυρκαγιές, τις δασικές πυρκαγιές και όλες τις καταστροφές, το να επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν υπάρχει κτηματολόγιο, ε, όπως ας πούμε γίνεται στην Ελλάδα, ε, αν δεν υπάρχει μια εθελοντική διαδικασία ε, για την πυρόσβεση, μια καλή αντιμετώπιση και πρόληψη των καταστροφών, δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα οργάνωσης. Αν κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε έναν παρεμβατισμό ευρωπαϊκό που θα εξελιχθεί. Θέλουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη από μόνα τους να λαμβάνουν τις ευθύνες. Οι πολίτες, οι πόλεις, ε, οι κοινότητες, ε, οι περιφέρειες και εμείς ε, να ερχόμαστε προσθετικά και να δίνουμε κονδύλια μέσα από τα περιφερειακά ταμεία. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν να υπάρχει στην έκθεση και ε, να επικεντρωθούμε στο θέμα ότι πρέπει να έχουμε βοήθεια για την αυτοβοήθεια και ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας την αρχή της επικορικότητας Και μόνο όταν ε, η τοπική δράση δεν φτάνει να μιλάμε για ευρωπαϊκή παρέμβαση. Όμως αυτό ε, να ε, γίνεται μόνο σε λίγα πράγματα όπου υπάρχει προστιθέμενη αξία από την Ευρωπαϊκή Παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Στα πλαίσια των κλιματολογικών αλλαγών χρειάζεται μια μακροπεριφερειακή προσέγγιση όπως έλεγε και ο κύριος Βλάσακ. Νομίζω λοιπόν ότι σε μια μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική που είναι απαραίτητη πρέπει να σκεφτούμε να δώσουμε κάποιον αυξημένο ρόλο στον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός ήταν πολύ, υπήρξε πολύ αποτελεσματικός για την αντιμετώπιση καταστροφών. Το 2011 είναι έτος εθελοντισμού και θα μπορούσαμε λοιπόν να τονίσουμε ιδιαίτερα την ε, σημασία που θα είχαν ομάδες εθελοντών και εθελοντριών και για την πρόληψη. Πρέπει να το κάνουμε, έτσι νομίζω. Very Mr. Kelly, you have the Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή ιδιαίτερα για τις πρακτικότατες συστάσεις του, ιδιαίτερα την νούμερο 5 που λέει ότι η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία. Ή μάλλον εκεί που λέει για την πρόληψη και το 5 όπου λέει ότι τα προγράμματα πρέπει να υποχρεωτικά να εμπεριέχουν κάποια αγγίηση πραγματικής τους εφαρμογής. Στη χώρα μου αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ότι ορισμένες ε, πόλεις που δεν είχαν σημειωθεί ποτέ πλημμύρες ε, χρειάστηκε και αυτές να εγκρίνουν προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιας περίπτωσης και αυτό είναι φρόνιμο. Αν είχαν υπάρξει τέτοια προγράμματα πρόληψης παντού νομίζω τα προβλήματα θα ήταν πολύ λιγότερα. Πρέπει λοιπόν οι εθνικές κυβερνήσεις να καταλάβουν ότι άμα δεν εφαρμόζουν τα πρότυπα δεν χρειάζεται καν, είναι μάταιο να έρχονται να χτυπάνε στην πόρτα, την πόρτα της Ένωσης για να ζητιανεύουν βοήθεια. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τον εισηγητή απόλυτα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. you have the floor, Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλφόνση. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι το ουσιώδες το οποίο δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Οι κίνδυνοι είναι ε, διαφορετικοί προς τη φύση του και στην ίδια πολιτική. Το να ε, παίρνουμε τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τους σεισμούς, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι συνετό. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα σεισμό, ε, σεισμό πάντα ε, θα δράσουμε κατόπιν της καταστροφής. Μπορούμε να προβλέψουμε κάποιες ισχυρές βροχοπτώσεις. Ε, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε τη βροχόπτωση. Εκεί λοιπόν η πρόληψη. Τώρα, ε, υπάρχουν ε, ε, σε άλλε περιπτώσει όμω μπορούμε να προβλέψουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να προβλέψουμε πότε και πού θα συμβεί μια καταστροφή σε ορισμένε περιπτώσει. Άρα, δρώντα προληπτικά, μπορούμε να αποφύγουμε όλε τι συνέπειε. Ενώ εκ των υστέρων βρισκόμαστε απέναντι σε καταστροφέ, σε τεράστιε καταστροφέ και στη φύση και στο περιβάλλον και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Παίρνω το παράδειγμα τη Κορσική, όπου έχουν γίνει πολλέ πυρκαγιέ. Για χρόνια δεν είχαμε ε, πυρκαγιές γιατί πραγματικά υπήρξε μια ε, πολιτική ε, να σβήνονται οι πυρκαγιές από την... μόλις, μόλις έχουμε μια σπίθα για παράδειγμα. Ε, με αυτόν τον τρόπο είχαμε τρομερά αποτελέσματα. Πέρσι όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο γιατί ξαφνικά οι μετεωρολογικές, οι συνθήκες ήταν ακραίες. Υπήρξαν βέβαια αεροπλάνα τα οποία παρενέβησαν αλλά τα μέσα των περιφερειών, τα μέσα των κρατών σε, σε περίπτωση ε, ακραίων καταστροφών δεν επαρκούν. Άρα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε η κοινότητα να διαθέτει μια τέτοια δύναμη που να παρεμβαίνει όταν, υπάρχουν τα, όταν ε, ε, έχουμε αυτές τις ακραίε περιπτώσεις. Έτσι ώστε να προλάβουν τα γεγονότα. Εγώ διαφωνώ λοιπόν με όσους πιστεύουν ότι ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να έχουμε ε, δυνάμεις παρέμβασης. Γιατί νομίζω ότι στις πυρκαγιές, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο. Thank Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να κάνω ορισμένα σύντομα σχόλια στα ελληνικά. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή για την εξαιρετική γνωμοδότηση. Περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές θέματος, τονίζοντας το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στον κύκλο διαχείρισης, καταστροφών, καθώς και τη σημασία της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση της πιθανότητας να βελτιωθεί η ένταξη της πρόληψης καταστροφών στα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί για την χρονική περίοδο 2007 έως και 2013. Θα μπορούσαμε ίσως να τονίσουμε επιπλέον την καθοριστική σημασία της γραμμής 112, ιδίως στο πλαίσιο των μέτρων ευαισθητοποίησης και προετοιμασίας των πολιτών. Δεύτερον, καθώς και το ρόλο του στόχου για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, ο οποίος μπορεί να είναι καθοριστικός για την διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειροτεχνίας και των πρακτικών στον τομέα πρόληψης των καταστροφών, καθώς και της δημιουργίας κοινών βάσεων δεδομένων και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ όμορων περιφερειών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντόιτς και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αφού ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά βεβαίως και τον εισηγητή. Κύριος Ντόιτς. <clears throat> Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω το εξή. Ε, όσον αφορά το θέμα αυτό, θα ήθελα να, να σας πω ότι ε, τα, τα γεγονότα, ε, τα πρόσφατα, μου άλλαξαν άποψη. Και επιτρέψτε μου, όσον αφορά το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης, να εκφράσω την επιθυμία μου η Επιτροπή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της γιατί ακριβώς ε, ε, είχαμε αυτά τα πρόσφατα γεγονότα στη Μαδέιρα. Υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Πάνω από 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την καταστροφή. και ε, ο σύντροφό μα, ο κύριο Τεσέρα, σήμερα το βράδυ δεν βρίσκεται εδώ γιατί έπρεπε να μεταβεί επιτόπου ε, στα πλαίσια τη προσπάθεια ε, να αντιμετωπιστούν οι συνέπειε αυτή τη καταστροφή. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό να λάβουμε όλη υπόψη αυτά τα γεγονότα. Γιατί ακριβώ πριν από λίγου μήνε μία αντιπροσωπεία της επιτροπή μα μετέβη στην Μαδέιρα για να γνωρίσει την κατάσταση ε, από πρώτο χέρι. Υπήρξε λοιπόν μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων, αλλά εκτό από την ανταλλαγή απόψεων αυτή τη στιγμή πρέπει να εκδηλώσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μα. Όχι μόνο στα λόγια, αν θέλετε, αλλά συγκεκριμένα. Και πρέπει να σα πω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει το δικό του ρόλο. Και ποιο είναι αυτό, να ε, ε, πούμε σε όλους αυτούς που υπέστησαν όλα αυτά τα τρομερά δεινά ότι είμαστε δίπλα τους και τους σκεφτόμαστε. Thank Σας ευχαριστώ. Ναι, ε, χαίρομαι ε, που είπατε αυτά, που είπατε γιατί ήμουν και πρόεδρος αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε την, ε, της Ματιμαδέρα και πραγματικά ε, λυπάμαι ιδιαίτερα για τα γεγονότα. Θα μεταφέρω το αίτημά σας και την επιθυμία σας στην κυρία Χούμπνερ για να ε, στείλουμε επιστολή που θα εκφράζουμε τη συμπάθειά μας και την αλληλεγγύη μας στα θύματα. Okay. like the... Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στην, ε, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Oui, merci, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, ευχαριστήσει την Επιτροπή σας και τον εισηγητή για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και για τη συμβολή σας στην έκθεση του κυρίου Φεραίρα για μια κοινοτική προσέγγιση της πρόληψης. Ευχαριστούμε επίσης γιατί υπογραμμίσατε το βασικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών ε, στον κύκλο διαχείρισης των, καταστροφών, δηλαδή πρόληψη, προετοιμασία, ανταπόκριση ε, και ανοικοδόμηση. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και θέλουμε να εργαστούμε με βάση τον κύκλο αυτό. Ε, αλληλεγγύη, ανταπόκριση, απάντηση, αλλά και περαιτέρω. Από την έγκριση της ανακοίνωσης αυτής το 2009 από τότε και στο μεταξύ χρονικό διάστημα ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υλοποιήσουμε αυτή την ανακοίνωση ε, σε επίπεδο εργασία, επί των βέλτιστων πρακτικών, επί τη ενημέρωση, ανάλυση κινδύνων, ε, χαρτογράφηση των κινδύνων και βεβαίω σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών που θα εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία και θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα το πιο συγκεκριμένο ερώτημα ε, των δημοσιονομικών πόρων, ξεκινήσαμε μία μελέτη για κριτική ανάλυση των ε, δημοσιονομικών μέσων στον τομέα τη πρόληψη και ελπίζουμε τα αποτελέσματα τη ανάλυση αυτή, τη μελέτη αυτή, να μα βοηθήσουν να εντάξουμε καλύτερα το στοιχείο ε, τη πρόληψη στα μέσα, τα δημοσιονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Εξάλλου, όπω πρότεινε και ο εισηγητή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ε, την ε, θέσπιση πιο άμεση σχέση ανάμεσα στο δημοσιονομικό μέσο και στην ε, εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως για παράδειγμα η πρόληψη των καταστροφών. Και εδώ, καταλαβαίνετε, εργαστούμε επί των μεθόδων, επί της μεθοδολογίας των διαδικασιών που θα μας επιτρέψουν τελικά μια αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των προβλέψεων ε, και θα έχουμε έτσι προσθέμενη αξία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, να σας ε, υπενθυμίσω ότι η 1η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι μπορεί να θεωρηθεί ε, η προθεσμία για την κατα έκθεση των τροπολογιών για να εγκριθεί τον Απρίλιο στην Ολομέλεια η έκθεση. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ε, να τονίσω ότι η Επιτροπή μας ε, δεν είναι η υπεύθυνη Επιτροπή, κύρια Επιτροπή για αυτό το θέμα. Εμείς απλά εξετάσαμε το έγγραφο, δεν θέλαμε να υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη με τις ιδέες που ήδη εκφράζονται. Όσον αφορά στην αλληλεγγύη, μια παρατήρηση. Φυσικά θα ληφθεί αυτό υπόψη, ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στη διεθνή ενίσχυση, το συντονισμό των δράσεων, ε, ε, επιμερισμό των ευθυνών, αλληλεγγύη κτλ. Όλοι οι συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στη γεωργία στο θέμα, ε, όσον αφορά στη διαχείριση των καταστροφών, γιατί η γεωργία ε, αποτελεί ένα μείζον ζήτημα και ε, χρηματοδοτείται από άλλα ταμεία, άλλες δομές και οι άλλες δομές ήδη προβλέπουν ενίσχυση στην γεωργία αρρωγή Επίσης, ε, θα λάβω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια και όταν θα είναι έτοιμο το τελικό κείμενο θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να συμπεριληφθούν. Okay, again, Ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση που κάναμε. Εφόσον δεν χρειάζεται να ληφθεί άλλη απόφαση από την Επιτροπή μας, ε, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής ε, Περιφερειακής Πολιτικής στην αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ειδικότερα ο στόχος 2. Η κυρία Ροδικράτση έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω στη διάθεση. Ε, μέγιστο μισή ώρα, κυρία Κράτση. Πόσο είπατε? Μισή ώρα. Στο για σύνολο. για όλο το ναι, θέμα. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να έχουμε τη δυνατότητα και συζήτησης. Ε, ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, με επιτρέπετε, να, ε, επειδή μιλάμε για την ε, πολιτική συνοχή σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπως είναι αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα στην Ευρώπη, ήθελα να υπενθυμίσω τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη γενικά, για τη σύγκληση που είναι στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων αλλά και για τον προγραμματισμό και τη στρατηγική μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής συνοχής ε, ε, σήμερα αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία λόγω του ότι ζούμε στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης με βαθιές επιπτώσεις των οποίων η, σημασία αναδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Ε, ένας λόγος παραπάνω είναι όχι μόνο η, ορατότητα των επιπτώσεων και η ανάγκη αντιμετώπισης τους, αλλά μια άλλη διαπίστωση ε, μας κάνει να στεκόμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο ρόλο που μπορεί να έχει η πολιτική συνοχής. Είναι ότι οι, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν έντονα τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των συνεπειών του στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στην παραγωγή, στη ζήτηση και στην απασχόληση και διότι παρατηρούμε ότι παρόλο την πολιτική ε, συνοχής, ακόμη και στην Ευρωζώνη έχουμε απόκληση των ανισοτήτων παρά σύγκληση. Και ορισμένες περιοχές πλήττονται ιδιαίτερα. Δεδομένου ότι έχουμε λίγα εργα... ένα χαμηλό κοινοτικό προϋπολογισμό που θα μπορούσε άμεσα να δώσει λύση σε προβλήματα της πραγματικής ε, οικονομίας. Με δεδομένο ότι έχουμε ασαφείς χαλαρούς μηχανισμούς αλληλεγγύης. Ε, αυτό που μας μένει είναι να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής με την ευρεία τους έννοια, δηλαδή τα διαρθρωτικά ταμεία και όλες τις άλλες πρωτοβουλίες και μέσα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των περιφερειών. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο που αποτελεί ένα ευρύτερο προβληματισμό που πιστεύω ότι πρέπει να, είναι, να γίνει και βασικός ε, προβληματισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς ε, εξετάζουμε το στόχο 2, τις περιοχές στο στόχο 2. Σας υπενθυμίζω ότι ο στόχος 2 έχει σκοπό, φυσικά όλοι γνωρίζουμε, να παρέμβει σε διαρθρωτικά προβλήματα στην πρώτη προγραμματική περίοδο 2000-2006 είχε να κάνει με τις περιοχές που είχαν καθυστέρηση στους αναπτυξιακούς δείκτες ε, και στις επιπτώσεις των αναπτυξιακών δικτών στην ε, οικονομία, στην έλλειψη κοινωνικής συνοχής, στις προβληματικές περιοχές όπως λέγαμε. Στην περίοδο την προγραμματική που διάγουμε τώρα, 2007-2013, ε, ο στόχος 2 αφορά καταρχάς τέσσερα περίπου εκατομμύρια κατοίκους και στοχεύει πιο συγκεκριμένα στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Στα κλειδιά δηλαδή της ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Ήδη μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πρώτης κρίσης έχουμε θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς τους αναπτυξιακούς. Και εκεί που έχουν πληγεί οι περιοχές της Ευρώπης όπως είναι οι βιομηχανικές περιοχές και εκεί παρατηρούμε ότι υπάρχει μια, υπήρχε μια στασιμότητα της επιβάρυνσης και όχι ε, ε, ύφεση. Λοιπόν, ως έστω και ας μην είναι ικανοποιητικά παντού τα αποτελέσματα, μπορούμε να διαπιστώσουμε την ε, θετική ε, παρέμβαση των, της πολιτικής συνοχής στις περιοχές του στόχου 2 θα μπορούσε να έχουμε περισσότερα συγκεντρωτικά και ποιοτικά στοιχεία, κάτι το οποίο λείπει από την αναζήτηση που έκανα. Χρειάζεται, πιστεύω, μια ειδική μελέτη, ακριβώς επειδή αποκτάει μια ιδιαίτερη σημασία λόγω των σημερινών καταστάσεων η παρέμβαση στο στόχο 2 και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ε, με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένω να δούμε και τις εκθέσεις που τα κράτη-μέλη οφείλουν να καταθέσουν, να υποβάλουν στο τέλος του 2009 και ελπίζω οι εκθέσεις αυτές να μην είναι απλά μια αποτύπωση στοιχείων, αλλά να περιλαμβάνουν και ποιοτικά στοιχεία και προτάσεις των κρατών μελών για την καλύτερη αξιοποίηση του στόχου 2 ε, οι παρεμβάσεις που μπορούσαμε εμείς να προτείνουμε εκ πρώτης όψεως είναι ε, καταρχάς, αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διευκολύνουμε τη χρησιμοποίηση των εργαλείων των, των διαθροτικών ταμείων. Ε, θα μπορούσε να, να δούμε πώς οι κανονισμοί θα είναι, ε, πόσο η, η διαχείριση θα μπορεί η διοικητική διαχείριση να πλουστευτεί ώστε να είναι προσβάσιμα πώς μπορούν να προωθηθούν μέτρα όπως είναι η προχρηματοδότηση ή η χρηματοδότηση 100% ε, για οικονομία χρόνου δεν θέλω να επεκταθώ πολύ, αλλά είναι ένα, πιστεύω ένα ε, ε, εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει πολλά κράτη που βρίσκονται σε δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, το να έχουν τη δυνατότητα του να χρηματοδοτήσουν ένα έργο που το θεωρούν προτεραιότητας και να μπορούν να το αποπληρώσουν στο πλαίσιο της προγραμματικής περίοδου. Ε, επίσης ε, πιστεύω ότι μπορούν από τα κράτη-μέλη ε, πια να αξιοποιηθούν καλύτερα, πιο έξυπνα, πιο αποτελεσματικά όλες οι ευκαιρίες που δίνονται από τα εργαλεία συνοχής για την πρόβλεψη των καταστάσεων. Να μην τρέχουμε μόνο πυροσβεστικά, να προβλέψουμε όπως ας πούμε οι κλιματικές αλλαγές αυτά που θα φέρουν τα καινούρια και να προσαρμόσουμε τα εργαλεία μας προς, προς τα εκεί. Απ' την άλλη πλευρά η, επιβάρυνση του κοινωνικού ε, ιστού ε, καλεί τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν ε, τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του εφικτού ε, σε ε, άμεσες προτεραιότητες που παρουσιάζονται ως συνέπειες της, της κρίσης. Μια άλλη πρόταση την οποία θα ήθελα να κάνω είναι ότι πρέπει με πολύ προσοχή να δούμε και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο το συντονισμό όλων των εργαλείων που έχουμε για την ε, ε, πολιτική συνοχή. Εκτός από τα διαφορετικά ταμεία πρέπει να δούμε ε, πώς θα αξιοποιήσουμε τα α, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ενέργειας, πώς θα έχουν οι περιοχές πρόσβαση σε αυτά. Είχα πάει πρόσφατα στην ε, ε, περιοχή της Εγνατίας στην πατρίδα μας, κύριε Πρόεδρε, και είδα πράγματι πώς μπορεί να αλλάξει η φυσιογνωμία όχι μόνο της ελληνικής ε, περιοχής της Υπήρου ε, και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ευρύτερα της Νότιας Ευρώπης, όταν στα διευρωπαϊκά δίκτυα υπάρχουν οι κατάλληλες προσβάσεις. Επίσης έχουμε άλλα εργαλεία, πρωτοβουλίες για την καινοτομία. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα πλαίσιο που προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση όπως είναι ο στόχος 2, να αξιοποιηθούν οι, οι ευκαιρίες για την καινοτομία, το έβδομο πλαίσιο για την έρευνα, είναι όταν πηγαίνουμε πιο κοντά στην πραγματική οικονομία, πιο πολύ στη ζώσα κατάσταση μιας περιοχής, αντιλαμβανόμαστε τις τεράστιες ε, δυνατότητες που έχουμε από την προσβασιμότητα στα εργαλεία και από το συντονισμό στην αξιοποίησή τους. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε σε γενικές γραμμές. Το έγγραφο που θα καταθέσω θα περιλαμβάνει και στατιστικά στοιχεία της σημερινής κατάστασης και ε, συγκριτικά με την εξέλιξη της ε, απόδοσης ε, της πολιτικής συνοχής στο στόχο 2 και φυσικά κάποιες προτάσεις. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω την την, ε, τις απόψεις των συναδέλφων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι πράγματι πρέπει να καταλάβουμε ότι κρούεται κόδωνα του κινδύνου με τα δημοσιονομικά προβλήματα που έχουν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τη δυσκολία μεγάλων επενδύσεων, τη δυσκολία χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, πόσο πρέπει περισσότερο από κάθε άλλη ε, ιστορική περίοδο να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και οι ευθύνε μου είναι το δεύτερο μήνυμα, είναι μοιρασμένε σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο και φυσικά σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Κράτσα για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μα είπετε. Dear colleagues, I'd Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας θυμίσω ότι το σχέδιο έκθεσης θα εξεταχθεί στις 17 Μαρτίου και όπως σας πληροφέσει η κυρία Κράτσα, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να στείλετε σχόλια Ενώ αυτή η συζήτηση σήμερα θεωρείται μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Επειδή πρέπει να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες στις 5, 5 και 10 έχουμε μόνο τέσσερι ε, ομιλητέ. Η κυρία Βέστιφαλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι για τη συνεργασία με την κυρία ε, Κράτσα και τις άλλες κοιόδες εισηγητές. Ε, θεωρίζω ότι αυτή η έκθεση μπορεί στην πράξη να είναι μια έκθεση η οποία θα βοηθήσει πολύ και θα έχει νόημα στην παρούσα κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά την κατάσταση των εργαζομένων στην Ευρώπη. Όλοι μας ανησυχούμε για τις ε, βαρύνουσες επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σχεδόν όλες οι περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης και τα κράτη πλήττονται. σε όλες, σε όλες τις χώρες. Για μας, τους σοσιαλδημοκράτες, η αντιμετώπιση της ε, κρίσης ε, είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως ε, τους εργαζομένους. Θέλουμε και πρέπει να καταφέρουμε να διατηρήσουμε όσο περισσότερες ε, θέσεις εργασίας γίνεται και να ξαναδημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για αυτές που χάθηκαν. Η ευρωπαϊκή η περιφερειακή πολιτική ε, έχει στη διάθεσή της την δυνατότητα δημιουργίας ε, περισσότερων και νέων θέσεων εργασίας, η οποία είναι μια βασική γραμμή της ε, περιφερειακής πολιτικής ε, για αυτή την περίοδο. Οι επιπτώσεις της κρίσης ε, στην οικονομία δεν πρέπει να οδηγήσουν στο να παρακλίνουμε από αυτές τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. Η υποστήριξη περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες, είναι πράγματα που και στην κρίση θα πρέπει να εφαρμοστούν με όλο μας το σθένος πρέπει ε, η ευρωπαϊκή πολιτική, η περιφερειακή πολιτική να έχει θετική συνεισφορά. Πριν την κρίση μπορούσαμε να δούμε ότι τα διαρθρωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πολλές περιφέρειες ε, κατάφεραν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είχαμε την περαιτέρω εκπαίδευση και την κατάρτιση και ε, προσπαθήσαμε να είναι οι περιφέρειες ε, ανεξάρτητες όσο γίνεται περισσότερο από τις βιομηχανίες. Τώρα θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε όσο γίνεται την κατάσταση από τις επιπτώσεις της κρίσης. Και γι' αυτό χρειάζεται ευελιξία στα διαρθρωτικά ε, ταμεία. Ακόμα και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα μέσα ε, προσαρμοσμένα στις τρέχουσες συνθήκες. Χαίρομαι και συντάσσομαι για αυτή την έκθεση και συντάσσομαι. Ευχαριστούμε κυρία Βέστφαλ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους άλλους χειόντες εισηγητές γιατί αυτό το θέμα της περιφερειακής ε, πολιτικής ε, για την πάταξη της οικονομικής κρίσης είναι ένα κεντρικό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μένα. Στην ανάλυση της οικονομικής κρίσης ε, διαπιστώνουμε ότι αρχικά αυτή η κρίση ήταν τραπεζική. Τα κράτη έδωσαν πολλά χρήματα και ο διεθνής τραπεζικό, για, να, για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τον διεθνή τραπεζικό κόσμο. Παρά από αυτά τα δισεκατομμύρια τώρα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις ζητούν πιστώσεις από τις τράπεζες και η κατάσταση είναι κρίσιμη, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ε, δύσκολα έχουν πρόσβαση σε δάνεια. Αυτό ε, θα μπορούσε να είναι και ένα κεντρικό κομμάτι της περιφερειακής ε, πολιτικής, δεύτερος στόχος, απασχόληση κτλ. Ε, ειδικότερα ε, βοήθεια σε επίπεδο ρευστοποίησης, βοήθεια για τη ρευστοποίηση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τη ρευστότητα, συγγνώμη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις συμπεριλάβουμε στις πολιτικές ενίσχυσης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επίσης ε, ανάγκη να μειώσουν τις ε, διαδικασίες έρευνας ε, που εκτελούν εξαιτίας προβλημάτων ρευστότητας και αυτό θα είναι πολύ κακό για τα μελλοντικά προϊόντα. Θεωρώ ότι η περιφερειακή στήριξη θα πρέπει να στηρίζει τη συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργασία με πανεπιστήμια έτσι ώστε ακόμα και στην κρίση να μπορέσει να συνεχιστεί η ερευνητική διαδικασία έτσι ώστε να υπάρχουν στο μέλλον τα κατάλληλα προϊόντα και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά είναι ε, στοιχεία ε, τα οποία επιδιώκει αυτή η έκθεση και θεωρώ ότι είναι καλό που σε αυτή την Επιτροπή συζητούμε αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία εισηγήτρια, όσον αφορά τη ε, συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Νομίζω ότι είναι ουσιώδες να επιμείνουμε στις συνέπειες της κρίσης αυτής ιδιαίτερα ε, ως προς τους πιο ευάλωτους ε, ε, πολίτες και σε που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Ενώ η στρατηγική της Λισαβόνας μιλούσε για εξάλληψη φτώχεια στην Ευρώπη, η κρίση θα ενισχύσει αντίθετα το φαινόμενο αυτό, όπως βλέπουμε και φέτος, με μια αύξηση της φτώχειας στα περισσότερα κράτη-μέλη. Άρα, οι περιοχές του στόχου 2 σίγουρα είναι οι περιοχές που θίγονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ε, ιδιαίτερα απαραίτητο να συνδεθούν ε, οι πόλεις σε αυτή την ε, προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης. Δηλαδή των δυσκολιών στην εξέβρεση εργασίας, στην εξέβρεση στέγης, τα προβλήματα εκπαίδευσης και υγείας και ε, στην ε, εγγύηση για την, οικονομική, για την κοινωνική στήριξη ε, των οικονομικών μέτρων. Οι, οι, οι ανισότητες ανάμεσα στις περιφέρειες δεν γεννήθηκε τώρα με την κρίση άλλωστε. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν μακροπρόθεσμα μέτρα κοινωνικής ε, υποστήριξης των οικονομικών μέτρων για ε, την ε, βιώσιμη ένταξη, συνεχιζόμενη ένταξη των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σαγκουράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος είναι δυνατό να είναι κανείς. Καταρχήν θα ήθελα να σημειώσω ότι ακόμα και πριν από την κρίση οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάθηκαν. Το σίγουρο είναι ότι με την κρίση αυτές οι ανισότητες θα ενταθούν ακόμα περισσότερο όσα χρήματα και αν ρίξουμε από το Ταμείο Συνοχής σε οποιοδήποτε ταμείο θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα συνασπισμό καπιταλιστικών χωρών και εδώ δρά απόλυτα ένα νόμο που λέει ανισόμετρη ανάπτυξη. Δεύτερον, όχι μόνο περιφέρειε, κύριε Πρόεδρε, ε, ε, αντιμετωπίζουν ανισότητε, τώρα έχουμε ολόκληρε χώρε. Σα ε, φέρνω μόνο το παράδειγμα τη χώρα μα, που όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αντιμετωπίζει την απειλή από χώρε άλλε να βρεθεί εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν συνάδει με τα κριτήρια σύμπληξη κτλ. Και ξέρετε το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω βεβαίως υπάρχουν και άλλες χώρες, αλλά θα έλεγα ότι και στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους λαούς και τους εργαζόμενους από Ρουμανία, Βουλγαρία ε, και Ουγγαρία, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο από ό,τι γνωρίζω. Και όταν γίνεται συζήτηση αν το χρέος της Ελλάδας θα το αναλάβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή δεν ξέρω εγώ ποιο, Καταλαβαίνετε κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα δεν είναι πια οι περιφέρειες. Κλείνω λέγοντας ότι θα έχει ενδιαφέρον η έκθεση, όμως ε, το θέμα είναι ότι όσο καιρό τα κριτήρια είναι ανταγωνιστικότητα και το κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων, τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν ταλαιπωρούν, δημιουργούν την ανεργία και τη φτώχεια, θα οξύνονται και θα γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αγκουράκη. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Κράτσα αν έχει ένα μικρό... Ε, ε, ε, επειδή ζήτησε ναι. το λόγο ο κύριο Νιστερόη, θα σας δώσω το λόγο, ναι, κυρία Κράτσα. Η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκφραστεί, κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν έχει ζητήσει το λόγο. Very short. Okay, Mr. Van uh, Nistelrooy, you have Thank the floor. Please try I, to be so yeah, brief. I will be. Κύριε το λόγο, παρακαλώ να είστε σύντομο. Ε, τη στιγμή που γίνεται αυτή η εργασία εδώ, υπάρχει και μια ειδική επιτροπή στο Κοινοβούλιο που ασχολείται με το θέμα τη κρίση, όπω ξέρετε. Η κυρία Χίπνερ δεν είναι εδώ, αλλά είναι και σε εκείνη την ε, επιτροπή και διασφαλίζει τη σχέση μεταξύ αυτού του θέματος και της εργασία μα Και θα ήθελα να τονίσω ότι τώρα που έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε αυτά τα δύο πράγματα είναι καλό. Η διαρθρωτική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική είναι μακροπρόθεσμη πολιτική και η κρίση, όπως είπε και ο κύριος Στόιρερ, έχει οδηγήσει ε, στο γεγονός ότι πολλές αστοχίες της ε, ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης πρέπει να αποκατασταθούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς η κρίση λειτουργεί στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης και τι σημαίνει για την πολιτική συνοχή μας και τα άλλα μέσα χρηματοδότησης. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε ερωτήματα κλειδιά και να φέρουμε και το θέμα της ε, εδαφικής συνοχής ε, στο τραπέζι. Ζητώ λοιπόν από την εισηγήτρια να συντονιστεί και με τις ε, συζητήσει στην άλλη επιτροπή, να υπάρχει μια σύνδεση και να έχουμε ένα ε, κείμενο το οποίο δεν θα είναι διαφορετικό, να έχουμε παρόμοια πράγματα στην Ολομέλεια. Κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες απόψεις τους. Συμμερίζομαι όλα αυτά που είπαν. Ε, είναι και στα δικό μου σκεπτικό η εδαφική συνοχή, να, να δειχθεί η σημασία της εδαφικής συνοχής. Ε, επίσης, ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μια παρένεση κλασικά κάνει το Κοινοβούλιο για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της κάθε περιφέρειας. Και επίσης το άλλο το οποίο συμμερίζομαι είναι ότι ε, το πρόβλημα που εξετάζουμε εντάσσεται σε ε, μια ευρύτερη ε, ικανότητα που πρέπει να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προώθησης της ισόρροπης ανάπτυξης. Όσο υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των χωρών, όσο δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα στη σύγκληση μεταξύ των χωρών, τόσο θα πλήττονται οι περιφέρειες και οι πληθυσμοί τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Εγώ ευχαριστώ κυρία Κράτσα. Ε,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 Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ε, καταρχάς, έχετε όλοι τις κάρτες σας. Παρακαλώ, μπορείτε να τις ε, εισαγάγετε στις ε, συσκευές για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Είστε όλοι έτοιμοι? Τότε ανοίγει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι? Και όλες. Τότε μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι μία φορά, αν γίνεται. Ο κύριος Κέλλη ψήφισε, άρα μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Okay, der... Φαίνεται ότι λειτουργεί το σύστημα. Περιμένουμε όμως μερικούς να φέρουν τις κάρτες τους. Ε, στο μεταξύ... Ε, να σας πω ότι η κυρία Κουνή θα πρέπει να ψηφίσει χωρίς ε, κάρτα. Είναι κάποιος άλλος που δεν έχει. Ξεκινάμε λοιπόν με την ε, σχέδιο γνωμοδότησης οργία ε, σε περιοχές ε, με φυσικά προβλήματα. Κυρία Φεραγκούτ, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? Κακτά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, καταπίπτουν οι 3, 4, 5, 6, 8. Ψηφίζουμε την 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν καταπίπτουν οι 11, 12, 13 και ψηφίζουμε την 14 η οποία ε, και, όπως και η 15 έχει αποσυρθεί άρα ψηφίζουμε την 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ α μάλλον καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε η 16 άρα ψηφίζουμε την 18 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα έχει και το στις κάρτες. Ε, ε, ξεκινάμε με την τροπολογία 19. Υπέρ κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για το σύνολο του εγγράφου. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 39 υπέρ, καμία κατά. Συγχαρητήρια. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία για το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών. Εισηγητής κ. Κέλλη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα χωριστή ψηφοφορία σε δύο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 Συγγνώμη. Μάλλον καταπίπτει. Α, α, όχι, η προηγούμενη απορρίφθηκε, άρα ξανά ψηφίζουμε την 8 κανονικά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 14 το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Μόνο το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Stimmen το πρώτο κομμάτι, 14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην τροπολογία της συμβαστική νούμερο 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει η 17 και η 19. Άρα ψηφίζουμε την 15. Για την 15 λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε λίγο αυτό. 18. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24 κατά, 18 υπέρ. Τώρα πάμε στην τροπολογία 20 σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Τροπολογία 21. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εγώ δεν ψήφισα, αλλά και εγώ θα την επέριπτα. 22, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έτσι καταπίπτουν οι 26 και 27. Τώρα ψηφίζουμε την 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε μία προφορική τροπολογία. Την βλέπετε εδώ στο έγγραφο. Ποιος είναι υπέρ, η κυρία Κρέλ. Συγγνώμη. Εμείς ε, ως ε, ομάδα είμαστε κατά της προφορικής. Το συζητήσαμε και πριν. Ε, μάλλον, ε, λοιπόν, καταπίπτει αυτή η προφορική τροπολογία. Ερχόμαστε στην 30. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 32 καταπίπτει, άρα πέφτουμε, ε, πηγαίνουμε στην 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 καταπίπτει Ψηφίζουμε την 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 36-37 καταπίπτουν, ψηφίζουμε την 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 42 ε, καταπίπτει εξαιτία τη υιοθέτηση τη τρο... συμβαστικής 3. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 36 υπέρ, 5 ψήφοι κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κέλλη.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 Ευχαριστούμε. Μπορούμε τώρα να πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να ζητήσω από το συνάδελφο να, που να πει δύο λόγια πριν από την ψηφοφορία. Α, ε, εκεί είσαστε, μάλιστα. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, βεβαίως, δεν μπορώ παρά να σας πω ότι αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για μένα, γιατί τη στιγμή που μιλώ εδώ, όπως γνωρίζετε, έγινε μια τρομερή καταστροφή στο νησί Μαδέιρα, στο νησί μου, και τώρα που σας μιλώ, πραγματικά... Ε, αποσύρουν διαρκώς ε, ε, πτώματα, 250 άτομα έχασαν την κατοικία τους, ε, δεκάδες τραυματίες, πάνω από 40 νεκροί όπως ξέρετε, άτομα τα οποία βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε πολύ δινή θέση, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, η ζώνη έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Καταλαβαίνετε γιατί τραγωδία μιλάμε. Ε, ε, δρόμοι, γέφυρες που έχουν εξαφανιστεί, σπίτια ολόκληρα που έχουν γκρεμιστεί και υπολογίζουν ότι βρίσκονται κάτω από τα ερήπια ακόμα πολύ θαμένοι, ε, κάτω από λάσπη, στο Φουντσάλ για παράδειγμα. Και δεν μπορώ παρά να σας τα πω όλα αυτά και βρίσκομαι εδώ αλλά αισθάνομαι απέραντι οδύνη απέναντι στα άτομα αυτά τα οποία επλήγησαν. Αισθάνομαι λοιπόν ιδιαίτερη λύπη και για τα θύματα και για τα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν την τύχη των οικείων τους. Για να επανέλθω λοιπόν στο ερώτημα αυτό, στο θέμα αυτό, σας ομολογώ ότι αυτό αποτελεί ε, τρομερή προσπάθεια για μένα. Βρίσκομαι εδώ με το σώμα μου αλλά και με το πνεύμα μου. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ήδη ε, τις προηγούμενες φορές είχα την ευκαιρία να ε, σας μιλήσω για τους λόγους του οποίου οποίους ε, υπέβαλα τροπολογία στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα στην ε, διαγραφή της 4 που είχα υποβάλει εγώ ίδιος μετά από επαφές με τις περιφερειακές αρχές αλλά και με την Επιτροπή που δέχτηκε τον κατάλογο των προϊόντων που είχαν υποβάλει τα κράτη-μέλη τη στιγμή της έγκρισης ε, των προγραμμάτων. Άρα λοιπόν αυτή η λύση, παρόλο που ήταν άτυπη, αποτελούσε μια λύση που μας βοηθούσε να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας, άρα θεώρησα ότι δεν είχε λόγο πλέον να υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη τροπολογία. Δεύτερη παρατήρηση. Όσον αφορά το συμπληρωματικό κείμενο στην ε, τροπολογία 5, χάρη στην προφορική τροπολογία που έχετε στον κατάλογο ψηφοφορίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, επικυροποιούνται ε, τακτικά οι μέγιστε ποσότητε και εξαγωγέ και εισαγωγέ των μεταπημένων προϊόντων. Γι' αυτό πρότεινα να στηριχθούμε στο μέσο όρο των τριών προηγουμένων ετών. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε το ελάχιστο όριο με βάση τα έτη 89-90-91, δηλαδή τα έτη αναφοράς του ε, υφιστάμενου κανονισμού. Επίσης, για να ε, έχουμε περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση των ποσοτήτων, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο ποσό που να λαμβάνονται υπόψη και οι κοινωτικέ χώρε και οι τρίτε χώρε. Και μετά από επαφέ με του συναδέλφου και με τι άκρω απομακρυσμένε περιφέρειες αποφάσισα να υποστηρίξω τις τροπολογίε που προστατεύουν τις ε, ε, περιφέρειες αυτές και τα συμφέροντά τους. και περιμένουμε βεβαίως την τροπολογία που του κανονισμού, την τροποποίηση του κανονισμού που ανακοίνωσε η Επιτροπή για τον Ιούνιο. Και βεβαίως... Ε, Έχουμε και τον κανονισμό 793 του 2006, γιατί συνδέονται άμεσα τα κείμενα αυτά και με άλλους κανονισμούς. Ευχαριστούμε κύριε Τεξέιρα και να πω το εξή. Όταν ε, δεν ήσασταν εδώ όταν συζητήσαμε το θέμα 6 ημερήσια διάταξη για τι ε, ε φυσικέ καταστροφέ. Εκεί συζητήσαμε και το θέμα τη Μαδέρα και πήραμε την απόφαση να στείλω επιστολή ε, προ αρχέ ε, ε, όπου να εκφράζουμε την οδύνη μας και να προσφέρουμε την συμπαράστασή μας και πόσο ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τον κανονισμό που θα ψηφίσουμε τώρα, από ό,τι κατάλαβα και η κυρία Γκρέσ θέλει να πάρει το λόγο ε, επί της προφορικής τροπολογίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, εκφράσω και εγώ ε, τη συμπαράστασή μου ε, προς ε, τους πολίτες του, της Μαδέρα. Τώρα όσον αφορά την προφορική τροπολογία, να υπενθυμίσω ότι ακόμα και αν η πρόταση που αφορά την συμπερίληψη του γάλακτος σε σκόνη στα γαλακτοκομικά προϊόντα, εδώ υπάρχει ο εξή κίνδυνος. Να χάσουμε το στόχο της αυτάρκειας, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η αυτάρκεια όμως είναι απολύτως απαραίτητη για πολλούς λόγους Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με θέματα πιστιστικής ασφάλειας και στη συνέχεια ε, ε, συνδέεται και με θέματα που αφορούν το κόστος και το περιβάλλον. Υπενθυμίζω ότι οι εισαγωγές στηρίζονται στη χρησιμοποίηση ενεργειακών πόρων και πετρελαϊκών πόρων όσον αφορά τις μεταφορές. Και καταλαβαίνετε ότι η τιμή θα αυξηθεί ε, ιδιαίτερα τα προσεχή χρόνια. Απλά και μόνο ήθελα να πιστεί την προσοχή σας στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα τώρα μπορούμε να αρχίσουμε τις προφορίες. Ξεκινάμε την τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Αποσύστηκε. Δέκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά χιλιάδες εγκρίνεται 11 υπέρ κατά χιλιάδες εγκρίνεται προφορική τροποποίηση υπέρ κατά χιλιάδες απορρίπτεται και δεν εγκρίνεται 12 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται τώρα για το σκεπτικό 5 7 τροπολογία 7 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 1 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται προς το 6α είναι 8 τροπολογία 8 υπέρ Τά, ποιες εγκρίνεται. Για το 7 η 9 υπέρ κατά yes, εγκρίνεται. Για το 7α νέο το 2, η 2, η 2 υπέρ κατά. κατά. Ποιες εγκρίνεται. Συνολική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχισε. Έληξε. 38 υπέρ, δύο εποχές. Καμία ψήφος κατά. Εγκρίθηκε. Μπορούμε και να σε χειροκροτήσουμε αν θέλουμε. Τώρα το σημείο 11 11 εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης του κυρίου Όλτριχ Βλάσακ. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, χες, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, χες, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά χες γκρίνεται νομίζω τέσσερα Προπολογία. τέσσερα υπέρ κατά πόχε το ε, πρώτο μέρος ήταν αυτό το δεύτερο υπέρ κατά αποχές κρίνεται τρία υπέρ κατά εποχές γκρίνεται τμήμα 3 τώρα η τροπολογία 5 που είχε πέσει, είχε αποσυρθεί 6 ε, υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 8 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 9 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 10 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 11 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 12 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 13 γλωσσική τροπολογία. Α, δεν την ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. 15. Δηλαδή, Περ. Κατά. Ποιε. Κρίνεται. 16 αποσύρθηκε. 17 έχει εκπέσει. 18. Υπέρ. 18. Κατά. Χε. Α, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Υπέρ, υπέρ. 19 υπέρ. Προφορική τροποποίηση είναι. Ναι, ναι, είπατε. Έτσι είπατε. Ναι. Ε, μάλιστα. Και τι κάνουμε με την προφορική, την ψηφίζουμε. Α, ε, ψηφίζουμε 19 υπέρ, ε, έχουμε ψηφίσει, έχουμε ψηφίσει. Είχατε δει, είχε εγκριθεί, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. 20 αποσύρθηκε, 21 υπέρ. Κατά. Βοχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η συνολική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Όχι ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Έχει ήδη αρχίσει. Μήπως ψήφισαν όλοι και όλε μπορούμε να ελίξουμε. λήξουμε. 40 ναι, ναι, υπέρ, μία ψήφο ε, κατά και καμία αποχή. Okay. Μήπως μπορούμε τώρα σύντομα να δούμε και το 12. Α, εσείς, ναι, ναι. Ολτρίτς. Θέλω στο τέλος της ψηφοφορίας να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές και συντονίστριες που κάνανε τη διαπραγμάτευση. Τελεία. Μάλιστα. Και εμείς σας ευχαριστούμε όλοι και όλες. Τώρα να περάσουμε σύντομα στο 12. Όπως ξέρετε η πρώτη συνάντηση για τις ομάδες εργασίας έγινε και λάβατε την αναφορά της γραμματείας για τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης συνάντησης. Δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε τώρα γιατί μας λείπει ο χρόνος. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα υπήρχε στην ε, ομάδα εργασίας αυτή το πρόγραμμα για το 2020 εκεί ο Βανίστελ Ρόι να μας πει σύντομα, σύντομα τι υπόθηκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Λοιπόν, εδώ ε, έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα το Ευρωπαϊκή Ένωση Στρατηγική 2020. Η στρατηγική που προτάθηκε για πρώτη διαβούλευση πέρυσι και τώρα θα συζητηθεί την Άνοιξη και μάλλον θα ξανασυζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφή τον Ιούνιο. Πρόκειται για ε, ένα, διάφορα σύνολα στρατηγικών και η εντύπωσή μας είναι τουλάχιστον ε, η εντύπωση των μελών της ομάδας ad hoc ότι πρέπει να είμαστε σε μία θέση όπου να μπορούμε να ασκήσουμε την επιρροή μας ε, στο συγκεκριμένο σημείο. Και με έκπληξή μας βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ε, δεν, ε, ότι εδώ, εδώ, δεν ακολουθείται η μεθοδολογία ότι να έχουμε μια βασική αρμόδια επιτροπή και τις άλλε που να συμβάλλουν. Και όμως είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Άρα, τι θέλω να πω ότι έχουμε την εντύπωση και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σε αυτή την εντύπωσή μου ότι πρώτον και ρωτώ θα ήταν δυνατόν ο πρόεδρος της Επιτροπής μας να αποστείλει ένα γράμμα ένα γράμμα πρόεδρο όπου να λέτε ότι για μας ε, το σωστό είναι να ακολουθεί η φυσιολογική, η συνηθισμένη διαδικασία του Κοινοβουλίου. Ίσως όχι το Μάρτιο, τουλάχιστον τον Ιούνιο. Δεύτερη ερώτηση. Θα κάνουμε συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, ε, πιθανά στη συνεδρίαση του Μαρτίου. Ρωτώ λοιπόν, είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και τρίτον, απευθύνουμε συντονιστές των άλλων ομάδων. Θα μπορούσαμε να δούμε, να ρίξουμε ματιά στην έκθεση Κώστας Λάσρα, του συναδέλφου από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, γιατί η έκθεση αυτή αναφέρεται στις αδίκες της Λισαβόνας. Και πιστεύω ότι θα ήταν δυνατόν ή εν λόγω έκθεση να εστιάσει την προσοχή της στατική 2020. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να φτιάξουμε μια γέφυρα ανάμεσα στη Λισαβόνα στρατηγικής Λισαβόνας και στρατηγική 2020 και έχω την εντύπωση ότι αυτό στη συνέχεια θα μπορούσε να πάει στην Ολομέλεια. Τρία θέματα λοιπόν τα οποία πιστεύουμε εμείς, όταν λέω εμείς εννοώ τα μέλη της ομάδας ad hoc που είμαστε μια ομάδα εργασία. Που βεβαίω δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο τη Επιτροπή, απλά και μόνο θέτω τα ζητήματα αυτά επιτάπητο. Και τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω με την άδειά σα είναι το εξή. Δεν υπάρχει πρόθεση για συζήτηση στι επιτροπέ, αλλά θα υπάρξει ένα ψήφισμα. Ψήφισμα πριν από την Ολομέλεια του Μαρτίου. Άρα, νομίζω ήταν καλό εάν διαμέσου πρωτοβουλία, με πρωτοβουλία των διαφόρων πολιτικών ομάδων, να ενημερώσουμε ένα τον άλλον και έτσι να ξέρουμε όλοι πού βρίσκονται διάφορε θέσει και ποιε είναι οι απόψει των πόλεων, των περιφερειών και να δούμε στην τελευταία ανάλυση πώς όλα αυτά θα μπορούν να ληφθούν υπόψη στα ψηφίσματα που θα προετοιμάσουν οι πολιτικέ ομάδε Στην αρχή αυτή τη εβδομάδα θα είμαι σε θέση να σας δώσω το κείμενο του ΕΛΚ. Είναι ένα κείμενο το οποίο δεν υποβάλλει συστάσει ή δεν δίνει συμβουλέ. Απλά και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση συζήτηση με τι υπόλοιπε ομάδε. Αυτό θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε. Και, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Λαμπέρ και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μα. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω το εξή. Σα ζητώ να συμφωνήσετε με την πρόταση αυτή ε, αποστολή επιστολών από την Πρόεδρο και στην ομάδα οίκων, ε, αλλά και, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και στη διάσκεψη των Προέδρων για να εκφράσουμε τις απόψεις μας και τον τρόπο τον οποίο ε, γίνεται ο χειρισμός αυτού του ζητήματος. Αλλά να δράσουμε και επικοδομητικά, να κάνουμε τη ζήτηση αυτή. Το δεύτερο, επειδή ο κύριος Κάστρο Λάσσα δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, θα ε, το συζητήσουμε μαζί του, θα συζητήσουμε αυτή την ιδέα μετατροπής της δικής του έκθεσης στην έκθεση που θα αναφέρεται και στην ε, στρατηγική 2020. Αν συμφωνήσουμε, τότε θα μπορούσαμε να κινηθούμε προ τα μπρο και το Μάρτιο να πάρουμε όλε τι αποφάσει. Στο μεταξύ, ε, ε, πιστεύω ότι οι συντονιστέ θα είναι σε θέση να συμφωνήσουν για το πώ θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Πάντω, σίγουρα θέλουμε να είμαστε δραστήριοι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Αυτό ήθελα να πω. Αυτή είναι η πρότασή μου, αν συμφωνείτε. Τότε, εντάξει, ωραία, κλείνει το σημείο αυτό. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα, Λαμπέρ, και πάμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Και ε, καλωσορίζω με όλη μου την καρδιά τον κύριο Φίλιπ Μάιστατ, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σα καλήσαμε, σας καλήσαμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα με αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή και Κοινωνική Συνοχή. Αξιολογούμε ιδιαίτερα εμεί ω Κοινοβούλιο αυτή την ιδέα ε, ανάμειξη ε, των πολιτικών δηλαδή θέματα οικονομικής μηχανικής να τα συνδέουμε με θέματα πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εν ώψη του μέλλοντος. Γι' αυτό η ανταλλαγή απόψεων μαζί σα σήμερα θα αποτελέσει για μας ένα ε, ένα πολύ ε, ε, μια πολύ χρήσιμη εμπειρία. Σας ζητώ λοιπόν να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή και στη συνέχεια να απαντήσετε σε ερωτήσεις ή σχόλια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μου είπαν ότι καλύτερα να μιλούσα στη μητρική μου γλώσσα. Αν όμω προτιμάτε μπορώ και στη γλώσσα του Σέξπιρ. Ποια είναι η εθνική σας γλώσσα, είναι τα γαλλικά αν και είμαι Βέλγος γιατί είμαι γαλλόφωνος Βέλγος φαίνεται. Αν όμως προτιμάτε, αν όμως προτιμάτε, Τέλο πάντων, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Ήδη είπατε ότι η ΕΤΕ συνεργάζεται στενά με την Κομισιόν και ιδιαίτερα με σας κυρία Πρόεδρέ μου και αυτό είναι φυσικό διότι η ΕΤΕ είναι διεθνής δημοσιονομικός οργανισμός και λειτουργεί σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Ρώμης. Έχει δηλαδή μια πολύ συγκεκριμένη εντολή να στηρίζει δημοσιονομικά χρηματικά την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα φυσικό είναι να έχει στενή συνεργασία και με άλλα χρηματο... και με άλλους, άλλους θεσμικούς φορείς της Ένωσης και μεταξύ των οποίων βέβαια και το Κοινοβούλιο. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν προσέρχομαι πάντοτε σε αυτό, όχι διότι με υποχρεώνουν, γιατί η συνθήκη δεν προβλέπει τίποτε ως προς τις σχέσεις μεταξύ ΕΤΕ και Κοινοβουλίου. Αλλά επειδή μου φαίνεται τελείως φυσικό το δημοσιονομικό εργαλείο της Ένωσης να κάνει απολογισμό συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα τώρα για την περιφερειακή πολιτική. Προφανώς είναι από τις προτεραιότητες της ΕΤΕ γιατί τα λέει ρητά η συνθήκη. Να, να σας διαβάσω εδώ τι λέει το 309 από τη Συνθήκη Λισαβόνα και μετά βέβαια. Λέει ρητά ότι η εντολή της ΕΤΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και προσθέτει επίσης ρητά, αν όχι ρητότερα, ότι αυτό πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ένωσης. Η ίδια η συνθήκη λοιπόν βλέπετε λέει ότι η ΕΤΕ πρέπει να συνεργάζεται με την Κομισιόν ιδιαίτερα ως προς τη χρήση των διαφορετικών ταμείων. Η χρηματοδότηση λοιπόν προγραμμάτων στις λεγόμενες περιφέρειες σύγκλησης είναι από τις προτεραιότητες της ΕΤΕ. Το 2009 χρηματοδοτήσαμε 205 προγράμματα στις περιοχές αυτές, συνολικού ύψους 29 δισεκατομμυρίων. Και επειδή πέρυσι υπογράψαμε δάνεια για 79 δισεκατομμύρια, η ΕΤΕ είναι Φαίνεται πως είναι ο πιο σημαντικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Ένωσης. Δεύτερος μόνο προς την Παγκόσμια Τράπεζα. Και αυτό το ποσό των 29 δισεκατομμυρίων για περιοχής σύγκλησης είναι 30% των δραστηριοτήτων μας και αύξηση κατά 38% του προηγούμενου έτους, έως προς το προηγούμενο έτος. Τα δάνεια αυτά είναι ισορροπημένα, με, κατανέμονται μεταξύ νέων και παλαιών χωρών μελών και μεταξύ χωρών μελών γενικότερα. Έχουμε χρηματοδοτήσει δάνεια σε ύψος 16 δισεκατομμυρίων για τις παλαιές χώρες και 13 για τις καινούργιες, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο στις νέες χώρες μέλη παρότι στις παλαιότερες. Να σας δείξω μερικά στοιχεία. Το ύψος των δανειοδοτήσεών μας είναι υψηλότερο στα μεγάλα κράτη βέβαια και γι' αυτό δεν είναι εκπληκτικό το ότι η χώρα που αποφελείται περισσότερο από τα δάνειά μας είναι η Ισπανία στις χώρες σύγκλησης ενώ με 4 δισεκατομμύρια και μισό και μετά αμέσως η Πολωνία 4 δισεκατομμύρια χιλιάδες. Φυσικό είναι λόγω της επιφανίας των χωρών αυτών. Με όρους όμως ανακεφαλήν, ανακάτοικο, τα στοιχεία αλλάζουν. Η Εσθονία τότε είναι η πρώτη. Αν τα υπολογίσουμε τα δάνειά μας ανακάτοικο. Η Εσθονία και μετά η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία. Ο ανατομέα τώρα πάνω από τα μισά δάνεια αυτά χορηγούνται για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και στις μεταφορές. Έχουμε όμως επίσης στηρίξει και προγράμματα και σε άλλους τομείς όπως στη λεγόμενη οικονομία της γνώσης, έρευνα, και ανάπτυξη και καινοτομία. Αν μου το επιτρέπετε λοιπόν κυρία Πρόεδρε θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ ιδιαίτερα σε μια καινοτομία των τελευταίων ετών, δηλαδή στενή συνεργασία μεταξύ Κομισιών και ΕΤΕ για τη χρήση των διαφορετικών ταμείων. Ένας τρόπος με τον οποίο στηρίζει η ΕΤΕ καλύτερη χρήση των διαφορετικών ταμείων είναι χρηματοδότηση του αντισταθμίσματος. Γιατί όπως ξέρετε τα κράτη που υποφελούνται από διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να κάνουν και μία δική τους συμβολή και τα έχουμε βοηθήσει στην εθνική αυτή τους συμβολή. Στη δική μας γλώσσα αυτά τα λέμε Structural Program Loans και τα χρησιμοποιήσαμε πέρυσι σε ύψος 3 δισεκατομμυρίων και πάνω. Αυτό είναι μια πολιτική συνεργασίας που επιτρέπει σε μερικές περιπτώσεις την επιτάχυνση της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων και για τις περιοχές της σύγκλησης. Ναι, πράγματι με χώρες μέλη για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στις περιφέρειες σύγκλησης. Αλλά όχι μόνον αυτό κυρία Πρόεδρε, διότι μαζί με σας Οργανώσαμε και πιο προωθημένες μορφές συνεργασίας. Θυμάμαι τον Απρίλιο του 2005 μια συνάντηση στο γραφείο σας όπου είχαν τεθεί οι βάσεις αυτής της συνεργασίας που μεταφράστηκε μετά στα λεγόμενα τέσσερα γάμα στη γλώσσα μας. Τζάσπερ, Τζέρεμι, Τζέσικα και Τζάσμιν. Τέσσερα j εδώ θα κάνω ένα σύντομο απολογισμό των τεσσάρων αυτών J ή J. Jaspers πρώτα. Είναι πρόγραμμα, κοινό πρόγραμμα της Κομισιόν της ΕΤΕ, της BERD και από το 2008 και της γερμανικής CAV, δηλαδή μια κοινή χρησιμοποίηση τεχνικών και άλλων μέσων για την προετοιμασία προγραμμάτων που μπορεί να χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι δηλαδή μέτρο για καλύτερη και γρηγορότερη χρησιμοποίηση των διαθροτικών ταμείων. Καλύτερη λοιπόν προετοιμασία των προγραμμάτων στις μεταφορές, των περιβάλλον, στην ενέργεια. Το 2009 μάλιστα 130 τέτοια προγράμματα προετοιμάστηκαν από το Jaspers 130 προγράμματα το 2009, κυρίως στην Πολωνία, την Τσεχία και τη Ρουμανία. Συνολικά 240 προγράμματα προετοιμάστηκαν από το Jaspers και διαπιστώνουμε ότι τα προγράμματα που προετοιμάστηκαν από το Jaspers έγιναν δεκτά πιο γρήγορα από την Κομισιόν για τη χορήγηση διαρθρωτικών κονδυλίων. Ιδιαίτερα όπως είπα και πριν στον τομέα του ύδατος είτε καθαρισμό είτε άλλες χρήσεις. 23% των προγραμμάτων που προετοίμασε το Τζάσπερς αφορούσαν το είδωρο αλλά και τις μεταφορές, λιμάνια, αερολιμένες και στην ενέργεια που είναι οι τρεις κύριοι τομείς που, με τους οποίους ασχολήθηκε το Τζάσπερς. Το δεύτερο γιώτα ο Ιερεμίας Πρόκειται εδώ για μια ιδέα καινούρια η οποία συνίσταται στο εξή. Στην προσπάθεια μετατροπή μέρου των διαρθρωτικών ταμείων που σε γενικέ γραμμέ χρησιμοποιούνται ε, άπαξ ω επιδότηση, δηλαδή one shot, να μετατραπούν λοιπόν σε χρηματοπιστωτικό, σε χρηματοοικονομικό μέσο ανανεώσιμο. Μέσο. Μην πρόκειται λοιπόν για μια πρώτη απόπειρα να προσπαθήσουμε να φροντίσουμε έτσι ώστε τα διευθυντικά ταμεία να χρησιμοποιηθούν με έναν τρόπο ε, που να ξεφύγουμε αυτό το άπαξ και να γίνεται επανειλημμένα. Η ιδέα λοιπόν ε, που βρίσκεται πίσω από αυτά είναι να δοθεί βοήθεια, ε, ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πιστώσεις και άρα να ε, εφαρμοστεί εκεί όπου απαιτείται και εκεί όπου υπάρχουν ανεπάρκειες και κενά να ε, ε, χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν χρηματοπιστωτικά, χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία βέβαια θα είναι ποικίλα ανάλογα με την, περιοφ... με περιφέρεια μερικές φορές θα πρόκειται για ταμείο εγγυήσεων άλλες περιπτώσεις θα πρόκειται για ταμείο συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλες φορές ε, οργανισμοί μικροπιστώσεων το θέμα εξαρτάται από την ανάλυση που θα γίνει σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιφέρεια με στόχο να καλυφθούν τα κενά και να εφαρμοστούν αυτά τα οικονομικά μέσα τα οποία λείπουν, χρηματοοικονομικά μέσα που λείπουν. Αυτό θα, αυτό, θα κάνει το Τζέρεμι. Μέχρι σήμερα 10 ταμεία Τζέρεμι έχουν υλοποιηθεί και συνολικό ποσό 1,8 ε, δις και ε, σε 7 κράτη-μέλη και σε 3 περιφέρειες. Τρίτον, το τρίτο Ζ είναι το Τζέσικα. Η ίδια ιδέα, ε, προσπάθεια λοιπόν χρησιμοποίηση των διευθυντικών ταμείων με έναν τρόπο που πάλι να έχουμε αυτόν τον ανανεώσιμο χαρακτήρα στον τομέα της ε, ανανέωσης των πόλεων. Να υπάρξουν λοιπόν χρήματα για την ανάπτυξη ε, την αστική. Κοινή προσπάθεια της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά εδώ ε, σε συνεργασία με την, με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ιδέα λοιπόν είναι να αφιερώσουμε μέρος των διαρθρωτικών ταμείων για την υλοποίηση ε, χρηματοοικονομικών μέσων, ταμείων δηλαδή αστικής ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 15 συμφωνίες επί της αρχής που έχουν υπογραφεί για δημιουργία δομών Τζέσικα σε μία σειρά από κράτη-μέλη και 8 ταμεία που ήδη έχουν ε, υλοποιηθεί για 900 ε, εκατομμύρια ευρώ. Και τέταρτον, το τελευταίο ζή είναι το Ζασμίν με στόχο την παροχή τεχνικής αρρωγής για την ανάπτυξη θεσμών μικροπιστώσεων. Προσθέτω εν συντομία, για να ολοκληρώσω την ε, εισαγωγή μου, ότι προσθέτω δύο άλλα μέσα κοινά Επιτροπή δηλαδή και ΕΠΕ γιατί μπορεί να μην αφορούν αποκλειστικά τις περιοχές σύγκλησης, αλλά ε, ε, συμπεριλαμβάνουν και αυτές. Το πρώτο είναι το ΕΛΕΝΑ, νέο μέσο χρηματοοικονομικής αρρωγής ε, από την Επιτροπή που διαχειρίζεται η ΕΠΕ, μέσω τεχνικής βοήθειας προς τις τοπικές αρχές, δήμους και κοινότητες, δηλαδή πόλεις, περιφέρειες, έτσι ώστε να υλοποιήσουν ερευνητικά προγράμματα στο τομέα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, των ανανεώσιμων ενεργειών και, της και των καθαρών μεταφορών είναι πρόσφατο, μόλις ξεκίνησε, αλλά ήδη διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αρκετέ αιτήσει εκ μέρου κυρίω των μεγάλων πόλεων που ζητούν βοήθεια για να μπορέσουν να υλοποιήσουν προγράμματα. Για παράδειγμα, συζητάμε τώρα με την πόλη των Παρισίων ένα πρόγραμμα ε, ανανέωση όλων των σχολείων ε, του Παρισιού ε, για ε, να υπάρχει ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αυτό θα γίνει και με πολλέ άλλε πόλει και εδώ έχουμε 15 εκατομμύρια ευρώ από την Επιτροπή για να ε, ε, παρέχεται αυτή η τεχνική και υποστήριξη για τα σχέδια αυτά, για τα έργα αυτά. Και τέλος, τελευταίο μέσο που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτό που ονομάζουμε ε, ε, sharing financial, risk sharing financial facility ε, για την έρευνα, δηλαδή χρηματοοικονομικό μέσο καταμερισμού του κινδύνου, του κινδύνου. Ξέρετε ότι τα ερευνητικά προγράμματα ποτέ δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι θα πετύχουν το στόχο τους αν δεν ολοκληρωθούν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κίνδυνο όσον αφορά τα ερευνητικά αυτά προγράμματα και μαζί με την Επιτροπή προσπαθήσαμε να βρούμε τα μέσα τα οποία θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, να αναλάβει περισσότερου κινδύνου στο συγκεκριμένο θέμα από ό,τι συνήθω. Συμφωνήσαμε λοιπόν στην εξή λύση. Δημιουργήσαμε ένα, ένα ε, ε, ε, ε προστατευτικού, δημιουργήσαμε ένα προστατευτικό μαξιλαράκι χρησιμοποιώντας ένα δις από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ένα δις από τα ετήσια κέρδη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δύο δις λοιπόν ευρώ, τα οποία θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε δάνεια πιο ε, ρηψοκίνδυνα αν θέλετε με αυτά που χρηματοδοτούμε συνήθως για ένα ποσό τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ. Ε, 10 ε, δις ευρώ. Ε, 10 εκατομμύρια, συγγνώμη. Ε, και μέσω αυτού του μέσου επιμερισμού του, ε, του κινδύνου. Το 2007 είχαμε ε, ένα ορισμένο ποσό, πέρυσι είχαμε ένα δις και ε, φέτος έχουμε τρία δις μέσω αυτού του κοινού μέσου. Κοινό μέσο, όπως σας είπα, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά θα σα αναφέρω εν είδη εισαγωγή και πιστεύω ότι ο διάλογο του το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τώρα θα προετοιμάσουμε ε, τι τις επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Από ό,τι άκουσα, η Επιτροπή σας θέλει να παρακολουθήσει από πολύ κοντά ε, την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Πράγματι, στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να σκεφτούμε τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους που θέτουμε. Και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι έτοιμη από, ε, να, να συμβάλλει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσει που θα μπορούσαν να εγκρίνουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με τι ερωτήσει και τα σχόλια. Ο Λάμπερ Βανίστερόι είναι ο πρώτο στο κατάλογο μου. Ευχαριστώ. Είναι μια πολύ καλή στιγμή για την πρόοδο που έγινε. Καταρχάς, ε, ποιος ε, εφήβρε όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα για τα προγράμματα. Ίδια άτομα εδώ. Σήμερα θα επιστρέψω στην Ολλανδία και θα πρέπει εκεί, επειδή έχουμε τις τοπικές εκλογές, να μιλήσω για το τι κάνουμε στην Ευρώπη. Θα μιλήσω για αυτές τις ε, ωραίες κυρίες και τα ονόματα που δώσανε. Ελένα. Σοβαρά τώρα. Μιλήσατε για το χρηματοδοτικό μέσο για την πρόληψη των κινδύνων. Ε, αν δούμε τώρα στην αγορά τι γίνεται με τις τράπεζες, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Παντού έχουμε κενά. Έχουμε ας πούμε κάπου τεχνολογικά πάρκα που πρέπει να γίνουν επενδύσεις με πανεπιστήμια κτλ. Μια τεράστια υποδομή που πρέπει να πληρωθεί και κανείς δεν μπαίνει σε αυτό. Ή θα μπουν σε 4-5 χρόνια. Αλλά θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη και αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε πιο εφευρετικοί ως προς τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε όταν ε, αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα προσπαθούμε να τα βάλουμε στην αγορά η Τζέσικα για παράδειγμα. Ποια είναι τα προβλήματα που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός του Κοινοβουλίου κτλ. κτλ. Ποια είναι, υπάρχουν. Γιατί θεωρώ ότι θα ήταν ενδιαφέρον ε, αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα που δημιουργήθηκαν, γεννήθηκαν πριν 3-4 χρόνια και στα οποία συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη τότε, φυσικά, Και θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη νέα γενιά καινοτόμων ε, χρηματοδοτικών μέσων και μέτρων τα επόμενα χρόνια ε, να δούμε τις επικρίσεις από την ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εκεί δεν υπάρχουν. όλοι χαίρονται με τα χρήματα που θα δοθούν στη Μόνικα και στη Τζέσικα. Ο κύριος Τρεμόπουλος έχει άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αυτός ο απολογισμός Okay. <clears throat> Ε, αυτός ο ε, για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι χρήσιμος και φανταζόμαστε θα υπάρχει πιο αναλυτικός και ίσως και έγγραφος εδώ για τα μέλη της Επιτροπής. Όμως <clears throat> θα ήθελα να μου πείτε, επειδή βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα ε, και έχει μεγάλη σημασία και με την πολιτική συνοχής αν θα ήθελα ένα σχόλιο για την κρίση που υπάρχει σε κάποιες χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μπορούσε ε, να κάνει κάτι για την έγκυρη αντιμετώπιση του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεύτερον επειδή εδώ συζητούσαμε και σήμερα για διάφορα λάθη που γίνονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων αν αυτά έχετε αντίστοιχη εμπειρία από τις δικές σας δραστηριότητες από τις διάφορες χώρες και σε τι ποσοστό μπορεί πίσω από τα λάθη να κρύβονται και απάτες. Έχουμε άλλου δύο ομιλητέ που ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Κράτσα πρώτα και η κυρία Ντέλη. Πρώτα η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω και εγώ τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αν θα μπορούσε πιο συγκεκριμένα να, μας, να αναφερθεί στη, στα, στους στόχους και στον απολογισμό των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Αυτό συνδέεται και με ένα θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως, την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε μια έκθεση στην οποία έχω την τιμή να είμαι συγκήτρια, για την πολιτική συνοχή και στο στόχο 2 την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Επειδή είναι το πρώτο ζητούμενο και ε, η αιτία πολλών θετικών προοπτικών για την ευρωπαϊκή οικονομία που ζητούμε η ανταγωνιστικότητα θα ήθελα ρωτήσω αν μπορείτε στο σημείο αυτό να κάνετε έναν απολογισμό μια αξιολόγηση των ε, δράσεων της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων και των προοπτικών που έχετε. σας ευχαριστώ. Ms. please. Κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Μιλήσατε για το ρόλο της ΕΤΕ στη χρηματοδότηση αστικής, ε, προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης. Όπως ξέρετε υπάρχουν πολύ σημαντικέ ανάγκε σήμερα για καθαρά κονδύλια και όχι δάνεια. Άρα, έχω απλή ερώτηση. Πώ μπορεί με τις τοπικές τα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συνεργαστεί η ΕΤΕ για να χρηματοδοτήσει όχι μόνο μεγάλα προγράμματα υποδομών, αλλά και μικρά προγράμματα και μέτρα βελτίωση ε, τη ενεργειακή αποδοτικότητας για τους κατοίκους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι ο κύριο ε, Φανίστερ Ρόι έθεσε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και θα πρέπει να το σκεφτούμε ειδικότερα στην ε, φάση υπερασκευής των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Ε, αντλήσαμε κάποια μαθήματα από το παρελθόν, φτιάξαμε κάποια καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, ανέφερα κάποια από αυτά, όμως είναι αλήθεια ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και δυσκολίες. Αναφέρατε και ο ίδιος μία από αυτές τις δυσκολίες. Οικονομικοί κανονισμοί, πάντοτε πρέπει να τους έχουμε υπόψη μας όταν φτιάχνουμε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για την πολυετή φύση των ε, προγραμμάτων. Δυστυχώς η Κομισιόν δεν μπορεί να δεσμευτεί για πάνω από ένα χρόνο. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε τέτοια χρηματοδοτικά μέσα αν δεν διασφαλίσουμε στους ε, ε, εταίρους μας ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον για μερικά χρόνια. Αυτό ο πολιτή χαρακτήρα λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να επιτρέπεται με του επόμενου κανονισμού. Φυσικά υπό όρους και υπό συνθήκες. Νομίζω όμως ότι έτσι σε κάποιες δικαιολογημένες περιπτώσεις θα έχουμε δικαιολογημένα τη δυνατότητα για πολιετή δέσμευση. Αυτά για τον ειδικό ε, κανονισμό για τα χρηματοδοτικά μέσα. Συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν. Όπως γνωρίζετε και όπως είπατε, δεν ακούσατε κανένα ε, παράπονο για το NSSF και ε, επειδή για το ΕΣΠΑ δηλαδή και αυτό είναι ένα πρόσφατο μέσο έχει γίνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση και θα πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτά για τους επόμενους ε, κανονισμούς. Ο κύριος Τρεμόπελος ε, έθεσε επίσης ένα τεράστιο θέμα για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης. Δεν θα μιλήσω τώρα εδώ για τον τρόπο που τα διάφορα κράτη-μέλη αντιδρούν. Να πω όμως ότι σύμφωνα με τα όσα έχουμε δύο ως τώρα γενικά, η αντίδραση των κρατών μελών ήταν πολύ καλή γιατί μπορέσαμε να ε, αποφύγουμε μια ύφεση πολύ μεγάλη, ακριβώ επειδή ε, η αντίδραση των κρατών μελών ήταν ε, διαφορετική. Η ταχεία αντίδραση των κρατών μελών με τα σχέδια ανάκαμψης έπαιξε συνολικά πολύ θετικό ρόλο. Αυτό σήμερα λοιπόν έχει ως ε, αποτέλεσμα Υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα στα περισσότερα κράτη-μέλη, όμως ήταν καλύτερη αυτή η γρήγορη αντίδραση των κρατών μελών παρά μια παθητικότητα που θα είχε πολύ πιο ε, σοβαρές συνέπειες. Φυσικά υπάρχουν ε, σφάλματα, δεν γνωρίζουμε τίποτα για απάτες, ε, όπως είπατε και εσείς και κάνατε και τη διάκριση. Όσον αφορά την ΕΤΕ, μας ζήτησαν μέσα στα πλαίσια αυτού του σχεδίου, του ευρωπαϊκού σχεδίου ε, για την ανάκαμψη της οικονομίας που εγκρίθηκε τον Δεκέμβρη του 2008 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητήθηκε από την ΕΤΕ να κάνει όσο πιο πολλά γίνεται και όσο πιο γρήγορα γίνεται για να αυξηθεί το, το μέγεθος των δανείων. Έτσι περάσαμε από τα 51 στα 79 δις, άρα πρόκειται για μια τεράστια αύξηση του όγκου των δανειοδοτήσεων και επίσης ε, ζητήθηκε αυτό να γίνει και σε τρεις κατευθύνσεις. Ε, πρώτον, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αύξηση δανειοδοτήσεων σε τράπεζες υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται αυτά τα ε, δάνεια για να βελτιωθούν οι συνθήκες πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης ε, για να δοθεί μια βεβαιότητα ότι τελικά όντως επωφελήθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν να θεωρήσαμε τους παραδοσιακούς τρόπους και περιλάβαμε αυτό το ε, νέο τύπο δανείων από τράπεζες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να μπορούμε να ε, επιβεβαιώσουμε ότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση την επέμβασή μας. Και αυτός ήταν ο πρώτος άξονας και πέρυσι μπορέσαμε να δανείσουμε πάνω από ε, σχεδόν 12 δις ε, για, στις τράπεζες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η χρήση είναι σχετικά γρήγορη. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο μας ζητήθηκε να επιμείνουμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη προτεραιότητα στις ε, περιφέρειες σύγκλησης, εκεί όπου η αύξηση των ε, δραστηριοτήτων μας ήταν μεγαλύτερη, για τις χώρες δηλαδή όπου υπάρχουν τέτοιες περιοχές ε, και τρίτον η ενέργεια στη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος. Αυτό εξηγεί ότι αυξήθηκαν ουσιαστικά τα δάνεια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω από 4 δις ε, δανείων πέρυσι για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για την αλλαγή του κλίματος, για την έρευνα σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, συγκεκριμένα για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, που εκπέμπουν τα μεταφορικά μέσα. δώστηκαν πολλά λοιπόν λεφτά σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με κινητήρες που θα, καταναλών, που θα εκπέμπουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, περιφέρειες σύγκλησης και μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος είναι οι προτεραιότητες που μας έδωσε το Συμβούλιο και ε, προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν οι πρόσθετες ενέργειές μας. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν υπάρχει και η ανησυχία που εξέφρασε η κυρία Κράτσα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, γι' αυτό τον λόγο προσπαθούμε να αυξήσουμε το μερίδιο των ε, δανείων που προσανατολίζονται στην οικονομία της γνώσης όπως ονομάζεται, την καινοτομία και την διάχυση νέων τεχνολογιών. Για να απαντήσω στην κυρία Ντελή, έχετε δίκιο, κυρία μου. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα πάντα με δάνεια. Πρέπει να υπάρχει και μια κεφαλαϊκή βάση και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της Τζέσικα. Με την Τζέσικα προσπαθούμε τα κράτη και οι περιφέρειες να επιλέγουν ένα κομμάτι των διαθωτικών ταμείων, το κονδυλίο που θα χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την ρευστότητα ή την ημιρευστότητα που θα χρηματοδοτήσει σε συνδυασμό με δάνεια τις ε, διαδικασίες ε, αστικής ανανέωσης. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που ακούστηκαν. Πράγματι τα 4 Ι, E, G, J στις ανατολικές χώρες και ιδιαίτερα στη δική μου τη Ρουμανία έπαιξαν πολύ επιτυχή ρόλο. Ήταν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το Jasper, ας πούμε μας επέτρεψε να εφαρμόσουμε πολύ σοβαρά προγράμματα για την ε, διανομή του ύδατος ας πούμε με μεγάλη επιτυχία. Και το ίδιο ισχύει και για άλλα προγράμματα τεχνικής υποβοήθησης. Την περασμένη εβδομάδα ήταν για μας πράσινη εβδομάδα. Και μας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Έλενα και καταλάβαμε και εμείς στη Ρουμανία πόσο σημαντικά είναι αυτά τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας τύπου Έλενας διότι πρόκειται για πολύ ενδιαφέροντες τομείς για το μέλλον, καθαρές μεταφορές, ενεργειακή αποτελεσματικότητα κλπ. Ερωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι τα ταμεία και άρα και τα 15 εκατομμύρια που προβλέπονται για μας θα μπορούσαν να συμπληρωθούν στο μέλλον λόγω του ενδιαφέροντος που έχουν αυτοί οι τομείς και από άλλα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Από την εμπειρία μου συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο Λαμπέρ. Ότι δηλαδή οι ισχύοντες διεθνείς κανόνες για τη χρηματοδότηση και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο υπήρξαν φραγμός πολλές φορές. Το ξέρουμε και από τα περασμένα χρόνια και τώρα που θα αρχίσουν να ισχύουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανονισμοί για την καινούργια περίοδο θα ήσασταν διατεθειμένος να συνεργαστείτε με την Κομισιόν στην αρχική τουλάχιστον φάση ώστε να απλοποιηθούν τα πράγματα περισσότερο και να μπορέσουμε και εμείς να συνδυάζουμε τα διάφορα ταμεία ευκολότερα και γρηγορότερα ιδίως στα πλαίσια της δημοσιονομικής κρίσης που μας πλήττει ώστε να δοθεί μια πρόσθετη όθηση. Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο, ξέρω. Ίσως να χρειαστεί χωριστός κανονισμός που να αναφέρεται ακριβώς στο θέμα αυτό του συνδυασμού των δημοσιονομικών εργαλείων. Δεύτερον, εσείς θα ήσασταν διατεθειμένος σε συνεργασία και με άλλους οργανισμούς στο μέλλον να αναλάβετε και περισσότερες δεσμεύσεις για τη χρήση του νέου αυτού εργαλείου ή θεωρείτε ότι τα προβλεφθέντα ήδη το εξαντλούν προς το παρόν τουλάχιστον τις δυνατότητες της τράπεζας δηλαδή ή μπορείτε εύκολα να προβλέψετε και επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών εφόσον μάλιστα ισχύει και η νέα συνθήκη και άρα δίνονται νέες δυνατότητες για τοπικές, για τοπικές πρωτοβουλίες όχι μόνο στο κεντρικό, εθνικό αλλά και στα περιφερειακά, τοπικά επίπεδα. Πώς το βλέπετε ως ρόλο της τράπεζας με βάση αυτές τις νέες τάσεις που παρατηρούνται. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα αυτά. Καταρχήν προς τον κύριο Ματούλα θα ήθελα να δηλώσω ότι επιβεβαιώνω αυτά που μας δήλωσε ότι στη Ρουμανία έχουν προετοιμαστεί πολύ σοβαρά και σημαντικά προγράμματα για το περιβάλλον ιδίως και την υγιεινότερη χρήση των υδάτων. Για την Έλενα που ρωτήσατε αν μπορούσαν να αυξηθούν τα κονδύλια της στο μέλλον και πέρα των 15 εκατομμυρίων, η Κομισιόν θα ήθελε να προτείνει περισσότερα, αλλά το θέμα είναι ο ενιάφσιος χαρακτήρ του προϋπολογισμού. Αλλά μπορείτε να είστε βέβαιος ότι θα ανανεωθούν τα προγράμματα και του χρόνου, όχι όμως από νομική σκοπιά. Δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα, πολιτική βεβαιότητα. Παραδείγματος χάρη χρειάζεται να δοθούν εγγυήσει για μακρύτερο χρονικό διάστημα από το ένα έτος αλλά που ακόμη δεν υπάρχουν λοιπόν. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το Έλενα στη Ρουμανία γιατί βλέπουμε τι τεράστιο ενδιαφέρον υπάρχει όχι μόνο στη Ρουμανία αλλά και για πόλεις ολόκληρης της Ένωσης. Τώρα κυρία Προεδρεύουσα ρωτήσατε αν μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα με τα προγράμματα Ι ή Μπορείτε να βασίσεστε στη συνεργασία μας, συνεχιζόμενη συνεργασία μας με την Κομισιόν για αυτά τα θέματα γιατί νομίζουμε ότι βοηθούν τα προγράμματα Ι στην επιτάχυνση της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων όλοι φαντάζομαι συμφωνείτε ότι το Τζάσπερ τουλάχιστον πρέπει να συνεχιστεί. Όσο για τον Ιερεμία και την Τζέσικα, αυτό είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι καινούριο και πιο δύσκολο να συνεχιστεί η εφαρμογή τους, αλλά, αλλά επειδή υπάρχουν θετικά προηγούμενα, υπάρχουν και αρνητικά αλλά πολλά πολύ καλά προηγούμενα, Νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα και από εκεί και να τα συνεχίσουμε και αυτά στην επόμενη δημοσιονομική χρήση αυτού του τύπου τα εργαλεία. Τέλος για το Τζάσμιν, για το Γιασεμί, ε, προς το παρόν συζητιέται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης να εφαρμοστεί μια νέα πρωτοβουλία μακροπίστωσης. Θα δούμε αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Διότι δεν είναι ούτε αυτή η πανάκια η μικροπίστωση. Αν θέλουμε όμως να φτάσουμε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουμε κάποιο εργαλείο για αυτές. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει μέχρι τις πιο μικρές επιχειρήσεις μικρότερες από τις μικρομεσαίες λεγόμενες ώστε να μπορέσουμε και τις μικρότατες αυτές επιχειρήσεις να στηρίξουμε με τεχνική υποβοήθηση μέσω του γιασεμιού αλλά και με άλλους τρόπους. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και σε αυτό πάντοτε και με τις υπηρεσίες της Κομισιόν για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ο Λαμπέρ. Να πούμε δύο λόγια για την νέα κατάσταση. Τώρα στο, το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται σε διαδικασία συναπόφαση, κυρίω όσον αφορά τα μέσα. Και ειλικρινά με εντυπωσιάζει το γεγονό ότι συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή κτλ. Αλλά νομίζω ότι σύντομα εμείς θα ξεκινήσουμε τις ακροασει. Για παράδειγμα, εμείς δική μας επιτροπή ε, τις ακροάσεις για, για το νέο ε, τρόπο σκέψης σε σχέση με τι συναπόφαση κτλ. Θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο να συμμετάσχετε και εσείς στην εργασία μας ευθύς εξ αρχή. Δηλαδή να συνεργάσετε στενά όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Κοινοβούλιο, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουμε αυξανόμενε ε, αρμοδιότητε εμεί στο Κοινοβούλιο σε αυτό το χρονικό διάστημα. σω λοιπόν έρθετε και στην ε, προσεχή ε, ακρόαση που θα διοργανώσουμε αυτό το χρόνο ω Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε μία πρόσκληση να συνεργαστείτε και με εμά ιδιαίτερα στενά. Ε, πράγματι, ε, ε, τώρα, εν ώψη των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, εμείς είμαστε σε ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο όσον αφορά όλους τους κανονισμούς Αυτό είναι αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Άρα, λοιπόν, ε, πρέπει να προετοιμάσουμε το μέλλον. Και μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι το κοινοβούλιο είναι πιο ανοιχτό στην καινοτομία, βεβαίως. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο δικό σας αυτό το, δεν είναι μόνο δική σας αυτή η εντύπωση. Το θέμα ε, έχει να κάνει βεβαίω και με την άμεση ευθύνη. Είμαστε λιγότερο άμεσα υπεύθυνοι, αν θέλετε, αλλά διευκολύνονται κάπω τα πράγματα. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσει και σχόλια, ε, θα ήθελα εξ ονόματο όλων μα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μάιστατ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήρθατε σήμερα στι Βρυξέλλε και ελπίζουμε να συνεργαστούμε πολύ πιο στενά στο μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ακόμα θέμα έχουμε στην ημερήσια διάταξη, οπότε μην φύγετε σας παρακαλώ.